Um, Καλημέρα σας συνάδελφοι, θα αρχίσουμε. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Πρώτη ανακοίνωση. Επαναλαμβάνεται, συνεχίζεται η διαθεσμική διαπραγμάτευση. 3 και 15 Σεπτεμβρίου αποφασίσαμε να επικυρώσουμε τους εισηγητές για τα επόμενα θέματα. Ευρωπόλ, Δίας Ντεμέρα, μεταφορά εμβάσματα από μαζί με την, αποκοινούμε την Επιτροπή Εικόνων για το ξέπλυμα βρωμίκου χρήματος η κυρία Σαρτζεντίνη κατά πολέμηση των απατών Λόπες Αγκυλάρ και οι επόμενοι τριμερείς διάλογοι θα αρχίσουν σύντομα για να γίνουν όπως πρέπει αυτές οι διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 75 του κανονισμού η Επιτροπή μας πρέπει να εγκρίνει όλα αυτά τα σχετικά νομοθετήματα με πλειοψηφία των μελών άμα τη ενάρξη των διαπραγματεύσεων. Αυτό θα καθορίσει βέβαια και τη σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας και όλα αυτά θα γνωστοποιούνται λέει το άρθρο 73 στον Πρόεδρο. Γι' αυτό προτείνω να συμπεράμε ένα νέο σημείο στην ημερήσια διάταξή μας, σύντομη παρουσίαση των εισηγητών για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τα τέσσερα αυτά μαθητήματα και προτείνω αυτό το πρόσθετο σημείο στις 5.30 το απόγευμα να το κάνουμε. Αν δεν έχετε αντιρρήσει, εγκρίνεται η, η σε διάταξη όπως τροποποιήθηκε. Υπάρχουν αντιρρήσεις μήπως. Τώρα ξυπνάτε βλέπω όλοι, άρα δεν έχετε αντιρρήσεις. Στο εξή όλες μας οι συνεδριάσεις θα γίνονται, θα αρχίζουν την ώρα που προβλέπετε. Δεύτερη ανακοίνωση, τα γλωσσικά. Η διερμηνία στα δανέζικα, λετονικά και κροατικά δεν υπάρχει. Στα μαλτέζικα δυστυχώς ούτε. Α, αρχίσει από τις 3 μέχρι τις 6 και συγγνώμη για τους ενδιαφερόμενους. Δεύτερον, το αίτημα των φιλελευθέρων για την Ουγγαρία. Έλαβα αίτημα των φιλελευθέρων για γραπτή ερώτηση προς την Κομισιόν σχετικά με τις παραβιάσεις των δημοσίων ελευθεριών και της ενόμου τάξεως στην Ουγγαρία. Της κυρίας μαζί με τον Λουί Μισελ, Ζαν Μαρί Καβαντά, Ζεράρ Ντεπρέ και Ναταλή Γκρίσμπεργκ επειδή η Κομισιόν δεν έχει δώσει γραπτή απάντηση στη διορία 6 εβδομάδων που προβλέπεται από τον κανονισμό 131 άρθρο αποφάσισα να φέρω το θέμα στην προσοχή σας ήρθα σε επαφή και με την Κομισιόν που υποσχέθηκε να δώσει τη γραπτή της απάντηση μέσα στην εβδομάδα όπως ξέρετε το θέμα των εξελίξεων στην Ουγγαρία ενδιαφέρει την Λίμπε και είναι στην ημερήσια διάταξη των συντονιστών αύριο προτείνω να τα συζητήσουμε εκεί στους συντονιστές ζητώ λοιπόν τους ρωτώ τους συναδέλφους αν συμφωνούν με την πρότασή μου αν έχουν αντιρρήσεις δεν έχουν τώρα μερικές από τις συστάσεις των συντονιστών και συντονιστριών για να τις εγκρίνουμε Πρώτον, η επιβεβαίωση των εισηγητών. Στη συνεδρία σήμερα στις 15 Ιουλίου οι συντονιστέ αποφάσισαν τι εξής δύο αρχές. Πρώτον, οι πρώην εισηγητέ που επανεξελέγησαν και είναι πάλι μέλη της Επιτροπής ΕΛΕΦ θα ξαναοριστούν. Το ίδιο είχαμε κάνει και στην προηγούμενη θητεία. Δεύτερον, Οι συντονιστές που όμως δεν είναι πια μέλη της ΕΛΕΦ πρέπει να, οι ομάδες που δεν έχουν τους ίδιους συντονιστές πρέπει να βρουν καινούριους, να ορίσουν καινούριους. Η δεύτερη αυτή αρχή σημαίνει ότι η κυρία Λούνατσεκ των Πράσινων αναλαμβάνει την οδηγία για την ίση μεταχείριση. Και ο ορισμός ηγητών για νέα νομοθετήματα, ορτεφέ, ορίζεται εισηγητής για τις θεωρήσεις και η κυρία Γκάλ του ΕΛΚ, εισηγήτρια για τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ΣΥΠΧΟ. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις εγκρίνονται όλα αυτά. Δεν υπάρχουν ούτε σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το σημείο 3. Η Κομισιόν θα μα παρουσιάσει τώρα την πέμπτη ετήσια έκθεσή τη για την Ανάστευση και το άσυλο. Παρέθεση 2013. Τα νέα μέλη μου είπαν ότι πριν έρθουμε εδώ στα, στην ουσία της διάταξη διάταξης πρέπει να εξηγήσουμε τα εξή. Οι εκθέσει για την κατάσταση που αφορά το άσυλο είναι έτοιμε από τον Ιούλιο και παρακαλώ τα νέα μέλη και να διαβάσουν το κείμενο που επισύω εδώ γιατί υπάρχει από τον Ιούλιο και σας δίνει την ευκαιρία να καταλάβετε τα προηγούμενα για να μπορείτε και εσείς να λάβετε μέρος στην συζήτηση για να καταλαβαίνετε και τι θα μας πει η Κομισιόν και τα λοιπά. Και τώρα καλώ την Κομισιόν να μας παρουσιάσει την πέμπτη ετήσια έκθεση της για τη μετανάστευση και το άσυλο 2013. Ορίστε κύριε Κοράδε Κυρία, κυρία. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Θα παρουσιάσω σύντομα τα βασικά σημεία της πέμπτης ετήσιας έκθεσης ε, για τη μετανάστευση και το άσυλο που εγκρίθηκε το Μάιο και μέχρι τώρα δεν είχαμε την ευκαιρία να την παρουσιάσουμε στην Επιτροπή σας. Αυτό, αυτή όπως ξέρετε η έκθεση δίνει μια γενική εικόνα των επιτευμάτων ε, στον τομέα της μετανάστευσης ε, και του ασύλου το 2013 καλύπτει και ζητήματα που αφορούν τη Βίζα και τη διοίκηση της Σέγγεν. Το 2013 γενικώ είδε πολλά επιτεύγματα όσον αφορά την οριστικοποίηση διαπραγματεύσεων σε πολλά νομοθετήματα, ειδικά στον τομέα της μετανάστευσης ασύλου και Σέγγεν. Ένα έτος που είχαμε επίσης αύξηση μεταναστευτικών ροών γενικώ και αιτήσεων ασύλου και είδαμε και προκλήσεις ε, όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές προς την Ένωση. Την 3η Οκτωβρίου, όπως ξέρατε, είχαμε τα τραγικά γεγονότα στη Λαμπεντούζα που οδήγησαν ε, την Κομισιόν ε, να φτιάξει μια ομάδα δράσεις ε, για τη Μεσόγειο και να βγάλει και μία ανακοίνωση το Δεκέμβριο για δράσεις που και μέτρα πρέπει να αναλυφθούν. Ο κύριος Σορίτ είχε μία συζήτηση με την Επιτροπή σας αρχές Σεπτεμβρίου για το θέμα αυτό, οπότε δεν θα επιμείνω, αλλά βεβαίως αν υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις, ευχαρίστως να απαντήσω όσον αφορά την νόμιμη μετανάστευση, τα βασικά επιτεύγματα οπωσδήποτε είναι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τους εποχικούς εργαζόμενους που ολοκληρώθηκε το 2013 ορίζονται κοινοί κανόνες όσον αφορά την εισδοχή και τα δικαιώματα αυτών των υπηκών τρίτων χωρών για να μην υπάρχει και εκμετάλλευση. Λίγο μετά, όχι εντός του 2013, αλλά καλό είναι να σας το πω, αρχές του 2014 ξεκινήσαμε και για τις ενδοετερικές ε, μεταθέσεις ε, ε, να διαπραγματευόμαστε την οδηγία για την εισδοχή δικαιώματα και κινητικότητα μετατιθέμενων ενδοετερικός. Τον Μάρτιο του 2013 η Κομισιόν υπέβαλε μία νέα πρόταση για οδηγία επαναδιατύπωσης για την υφιστάμενη ε, οδηγία ερευνητών και φοιτητών και για το πώς αναζητήσουν δουλειά αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, κινητικότητα εντός της Ένωσης, ειδικά για όσους υποφελούνται από προγράμματα όπως το Erasmus Plus το Marie Curie για ερευνητές κτλ. Και επίσης ε, προσπαθούμε να αναρμονίσουμε... και τους κανόνες για επικούς τρίτων χωρών που δεν ε, καλύπτονται ε, από υποχρεωτικούς ε, κανόνες για εκπαιδευόμενους υποαμοιβόμενους και τα λοιπά. Και ελπίζουμε να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις μόλις ολοκληρώσει και το Συμβούλιο την κοινή του προσέγγιση. Όπως ξέρετε το Κοινοβούλιο ε, τα έχει εγκρίνει ένα κείμενο στην πρώτη ανάγνωση και ελπίζουμε σύντομα να ολοκληρώσουμε. Το Δεκέμβριο του 2003 ετέθη ενισχύ η οδηγία για την ενιαία άδεια που καλύπτει έτσι και την απλοποίηση των διαδικασιών και τα δικαιώματα των υπηκών τρίτων χωρών που έρχονται για να εργαστούν και το καθεστώς των οποίων δεν ρυθμίζεται από τις νομιακές οδηγίες που αναφέραμε. Όπως παραδείγματος χάρη μπλε κάρτες, ε, εποχιακούς κτλ. Επίσης ε, συνεχίσαμε την παρακολούθηση της εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας και αυτό οδήγησε σε υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών ε, που κωδικοποιούν την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και δίνουν κάποιες οδηγίες για το πώς θα ερμηνευτεί η οδηγία. Επίσης, συνεχίσαμε τις προσπάθειές μας για την ενσωμάτωση. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει το δικαίωμα βεβαίως να περάσει ή να προτείνει νομοθεσία στο εθνικό επίπεδο αλλά χρηματοδοτούσαμε διάφορα έργα μέσα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ενσωμάτωσης, ε, ε, τους δείκτες ενσωμάτωσης ε, και τα εθνικά σημεία επαφών και το site μας. Το 2013 κάνουμε μια προσπάθεια να συμπεριληφθούν συστάσεις που αφορούν ειδικά τη μετανάστευση στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου όπου για κάποια κράτη-μέλη έχουμε στοχευμένες συστάσεις για την καλύτερη ενσωμάτωση υπηκών τρίτων χωρών, ειδικά όσον αφορά την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. Και θα συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον. Όσον αφορά το άσυλο και τη διεθνή προστασία, βασικό επίδευμα ήταν η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων του πακέτου προτάσεων ε, και την αναδιατύπωση του κανονισμού Eurodac για να υπάρχει ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου το οποίο τώρα πρέπει να εφαρμοστεί. Δεν θα αναφέρω την επιχειρησιακή πλευρά των δραστηριοτήτων αυτών. Θα τα πει αυτά ο κύριος Φίσερ. και οπωσδήποτε θα σφίτσει λεπτομέρειε. Όσον αφορά τώρα παράτυπη μετανάστευση, είχαμε νέες συμφωνίες επανεισδοχής ε, που υπογράφηκαν με τρίτες χώρες, ειδικά με την Αρμενία, Τουρκία και το Πράσινο Ακροτήριο. Συνεχίζουμε την, την ε, παρακολούθηση της εφαρμογής ε, της επιστροφής από τα κράτη-μέλη και ευθύσαμε και μία ανακοίνωση για τις επιστροφές και επίσης ε, αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε ένα εγχειρίδιο επιστροφών. Επίσης συνεχίζουμε την παρακολούθηση της οδηγίας κυρώσεων προς τους εργοδότες ε, όσων ε, απασχολούν ε, παρατύπως διαμένοντες μετανάστες και είπαμε στα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν τον κίνδυνο, να κάνουν επιθεωρήσεις, κάτι το οποίο έκαναν όλα τα κράτη-μέλη και αυτή τη στιγμή αξιολογούμε. Όσον αφορά την διαχείριση των συνόρων, η πίεση είναι ψηλή σε όλα τα εξωτερικά σύνορα. Η Frontex συνεχίζει τις δραστηριότητές της με κοινέ επιχειρήσεις στα εξωτερικά σύνορα. Ο κανονισμός Eurosur για την επιτήρηση των συνόρων ετέθη ισχύ το Δεκέμβριο του 2013 και ε, στοχεύει στην ε, καλύτερη παρακολούθηση διασυνοριακών εγκλημάτων και επιτήρηση και διάσωση εν πλώ. Επίσης, μετά από τις δύσκολες διαπραγματεύσεις για τη ε, διαχείριση του Σέγγεν, είχαμε ένα σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται. Είχαμε και την παρουσίαση του 2013 του πακέτου έξυπνων συνόρων που συμπεριλαμβάνει ένα σύστημα εισόδου-εξόδου και καταγεγραμμένων ταξιδιωτών και επίσης καταλήξαμε σε μια συμφωνία το 2013 για έναν μηχανισμό αμοιβαιότητας και άρσης ε, βίζας. Και τέλος, για να τελειώσουμε με τη βίζα, αρχές του 2013 παρουσιάσαμε και μια πρόταση για αναδιατύπωση του ε, κανονισμού βίζας. Όσον αφορά τη διεθνή διάσταση, ξέρετε πως το πλαίσιο ε, είναι η λεγόμενη συνολική προσέγγιση για την μετανάστευση και την κινητικότητα και βεβαίως έχουν συνεχιστεί οι δράσεις σε αυτόν τον τομέα να τονίσω ιδιαίτερα της Συμφωνίας Κινητικότητας με το Μαρόκο και το Αζερβαϊτζάν που υπογράφηκαν το 2013 και επίσης και τη συμφωνία με την Τινησία αρχές 2014. Επίσης, όσον αφορά τη σχέση με την ανάπτυξη. Ο διάλογος υψηλού επίπεδου του ΟΗΕ που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2013, στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισέφερε και συγκεκριμένα εγκρίναμε μία ανακοίνωση η οποία πλέον ενσωματώνεται πλήρως και στην αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015 τέλος Κάτι άλλο σημαντικό είναι πως το 2013 είχαμε και την πολιτική συμφωνία για το νέο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και την ε, σύσταση του νέου ταμείου μαζί με το Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας ε, το οποίο εγκρίθηκε αρχές του 2014 και είχαμε άρα τα πρώτα αυτά μέσα όσον αφορά άσυλο, μετανάστευση, επιστροφές και ενσωμάτωση. Θα τα βρείτε όλα αυτά στην έκθεση και στο έγγραφο εργασίας που περιέχει πιο λεπτομερείς εξηγήσεις της πρόοδου που έχει σημειωθεί, καθώς και ένα στατιστικό παράρτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κοράντο. Καλύψατε και, το άστυλο ε, και τη μετανάστευση. Δεν ξέρω αν ο Στίβεν Ράιαν θέλει να προσθέσει κάτι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται, διότι καλύψατε και τα θέματα σύλλου. Θέλετε να προσθέσετε κάτι, Στίβεν. Αν υπάρχουν ερωτήσεις ε, συγκεκριμένα θα απαντήσει ο Στίβεν. Ε, τα σχόλιά σας ε, στράφηκαν περισσότερο στη μετανάστευση, διότι μας ενδιαφέρουν και περισσότερο. Υπάρχουν πολλά πράγματα βέβαια να δούμε και για το άσυλο. Συνάδελφοι, αν έχετε διαβάσει βέβαια την έκθεση, μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις ε, και για το άσυλο και για τη μετανάστευση και οι δυο μπορείτε να απαντήσετε στη συνέχεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας δώσω το λόγο λοιπόν. Προφανώς ε, υπάρχει πολύ σημαντική δουλειά και στις δύο πτυχές και θέμα θέματα μετανάστευσης και θέματα ασύλου το 2013 και για τους συνάδελφους που μόλις ήρθαν ε, σας είπα ότι η έκθεση έχει δημοσιευθεί από τον Ιούλιο, παρά το γεγονός ότι συζητάτε σήμερα. Θα ξεκινήσει η συζήτηση, έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Σήμερα λοιπόν μπορείτε να πάρετε το χρόνο σας ε, και να σχολιάσετε και να θέσετε ερωτήσει. Μην το παρακάνετε όμως. Ε, η κυρία Σύπχολ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά. Ναι, ναι, ναι. είναι σαφές νομίζω τουλάχιστον μετά τα γεγονότα του Ιράκ και της Συρίας πως ε, στο προσεχές διάστημα θα αυξηθεί ο αριθμός των προσφύγων ε, ο αριθμός των προσφύγων οι οποίοι θα μπορούν να υποβάλουν μια αίτηση ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ όμως θέλω να θέσω ένα άλλο ερώτημα που αφορά την νόμιμη μετανάστευση. Η συνάλφουσα την Κομισιόν ανέφερε κάποιες πτυχές όπως ε, την οδηγία για εποχιακούς εργαζόμενους. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω το εάν η Κομισιόν ε, ε, έχει λάβει υπόψη τις άλλες δυνατότητες της νόμιμης μετανάστευσης. Δεν διάβασα ολόκληρη την έκθεση, οπότε θέλω να σας ρωτήσω εάν εξετάσατε στη, εάν εξετάσατε από τους πολλούς που προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη ε, και οι οποίοι δεν ε, μπορούν να υποβάλουν έτσι ασύλου εάν αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν ότι υπάρχουν και νόμιμοι τρόποι να έρθουν αν μπορείτε να με διαφωτίσετε ως προς αυτό και βεβαίως με ποιο τρόπο βεβαίως μπορούμε να ανοίξουμε και άλλους τρόπους νόμιμης μετανάστευσης Thanks, I think Ms. mentioned students and researchers and some other but Ευχαριστώ. Υπάρχουν και άλλες φαντάζομαι ερωτήσεις, αλλά θα σας απαντήσει στη συνέχεια. Ο κύριος ε, Κέρκο. Τι το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εν ώψη και της παρουσίασης που θα έχουμε λίγο αργότερα ε, φαντάζομαι ότι θα γίνει ένας χωρισμός ε, στο χρονοδιάγραμμα θα ήθελα να δω τι γίνεται με τα ε, πρότυπα για τις αιτήσει εσύλου στα κρατη μελου Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, κυρίως για το τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη και θα το θέσω αργότερα. Ε, όσον αφορά όμως το συγκεκριμένο ζήτημα, ναι, όντως ε, διατίθεται η έκθεση εδώ και αρκετό καιρό και είμαι βέβαιος ότι αρκετοί το διάβασαν στις καλοκαιρινές τις διακοπές ε, το κείμενο, αλλά επανεξετάζοντας το αυτό, ε, βλέπω ότι επισημαίνονται κάποια στοιχεία τα οποία με ανησυχούν ιδιαίτερα. Υπάρχει μνήμα στη Λαμπεντούζα φυσικά, υπάρχει μνήμα στην πολιτική, αλλά αυτά δεν συνέβησαν σε πολιτικό κενό. Με όλο το σεβασμό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους όσους εμπλέκονται, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της πολιτικής που έχει ένα πολύ μεγάλο κενό και αυτό είναι η πολιτική που εφαρμόζουμε για τα κράτη ή για τους οργανισμούς ή τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τον πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών που κατευθύνονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, συνήθως με ψευδείς ε, ε, δηλώσεις αντί να έρχονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι πραγματικά θέλουν να κάνουν αίτηση και να ενταχθούν στους κόλπου τη Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των κανόνων μετανάστευσής μας. Ε, θα πρέπει κάπω να είναι υπόλογε αυτέ οι χώρε που επιτρέπουν σε τόσο μεγάλο αριθμό ε, πολιτών του να φτάσουν ε, στις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλέ φορέ πρόκειται για εγκληματίες που εκβιάζουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους και παίρνουν μεγάλα ποσά για να φτάσουν εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ορισμένε από αυτές τις χώρες λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, είτε έμεσα είτε άμεσα, μέσω διαφόρων προγραμμάτων και αυτό φυσικά κάπως πρέπει να επανεξεταστεί. Οι χώρες αυτές δεν μπορούν να μην τιμωρούνται. Και επίσης, ε, Υποστηρίζουμε να υπάρχουν κατάλληλοι πόροι για το Frontex, ε, κατάλληλοι πόροι για τις ε, χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη αυτή τη στιγμή λόγω της γεωγραφικής τους θέσης αλλά δεν πιστεύω, και αυτό είναι κάτι το οποίο ίσως ε, ε, συζητάτε και σήμερα στη Χάγη, ε, στις συζητήσεις στην αστυνομία, στη Europol, θα πρέπει όμως να γίνει κάτι περισσότερο για να αντιμετωπίσουμε την, το διεθνές έγκλημα το οποίο μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση. Και δεν θα πρέπει να λησμονούμε, και με αυτό ολοκληρώνω, ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και κάποιες χώρες ε, αποτελούν δυναμίτη πραγματικά από πολιτική σκοπιά, διότι η πολιτική ε, είναι υπόλογη ενώπιον αυτών που αντιπροσωπεύουν και αυτοί που τους αντιπροσωπεύουν πιστεύουν ότι δεν συμπεριφερόμαστε με υπεύθυνο τρόπο και λογικό τρόπο. Θεωρούν ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε κρίση ε, υπάρχουν ε, ε, δηλώσεις για πολύ αυξημένο αριθμό ανθρώπων που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τονίζεται επίσης και ο αριθμός των ανθρώπων που χάνονται στη θάλασσα στην απέλπιδα προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ό,τι ανθρωπιστικά μέτρα και να εφαρμόσουμε, οτιδήποτε και αν δώσουμε, κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να είναι υπόλογος για αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν και εδώ νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα θεσμικά μας όργανα στην Ευρώπη θα πρέπει να ε, ιεραρχήσουν λίγο καλύτερα τις προτεραιότητές τους. Ιδάλλως, αν απλώς λέμε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εντάξουμε αυτούς τους ανθρώπους, δεν απαντάμε στο ερώτημα όσον αφορά τον αριθμό των ανθρώπων και τις κατηγορίες των ανθρώπων και των εγκληματιών που βρίσκονται πίσω από αυτές τις ε, δράσεις και τις χώρες που είναι υπεύθυνε. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό. Και Τέλος, για τα παιδιά. Θα ήθελα να αναφερθώ και λίγο στα παιδιά. Είμαστε στον 21ο αιώνα, τα πάντα είναι πολύ προηγμένα. Έχουμε τους υπολογιστές μας, ε, λογαριασμούς στο Twitter ε, ε, και σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαίνεται να μην εκτιμούμε το γεγονός ότι εξακολουθούμε να επιτρέπουμε να υπάρχει τεράστιος πόνος και ανήθικη συμπεριφορά ενώπιον παιδιών παιδιών ε, τα οποία πολλές φορές τα εκμεταλλεύονται ε, κλιματικά στοιχεία για ε, πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένες φορές αποτελούν το δόλωμα για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και πολλές φορές αυτά τα παιδιά στέλνονται σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ακόμα δεν έχουμε αρχίσει να ασχολούμαστε με κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει πουθενά τον 21ο αιώνα. Και μάλιστα όχι σε μία αναπτυγμένη και προηγμένη ε, περιοχή όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Τίμωθη. Ο κύριος Νίδερμιλερ. προηγμενη περιοχη οπως πολύ, κύριε κυριος Μιλλερ. ευχαριστω πολυ Επιτρέψτε μου να κάνω κάποια σχόλια για αυτή την έκθεση, στα ουγγρικά, αν μου επιτρέπετε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντική και κρίσιμη η συγκεκριμένη έκθεση και πιστεύω ότι συχνά δεν είμαστε αρκετά επιχρητικοί και δεν διαφοροποιούμε αρκετά ε, τις απόψεις μας. Πολλό δε μάλλον όταν αναφερόμαστε στην Ουγγαρία. Θεωρώ ότι η πολιτική ασύλου στην Ουγγαρία είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Πολύ πιο περιορισμένη από οπουδήποτε αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χωρίς υπερβολές νομίζω ότι δεν υπάρχει βιώσιμο σύστημα ασύλου στην Ουγγαρία αυτή τη στιγμή και υπάρχουν σχετικές δηλώσεις από πολλές ε, διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες και το 2013 δόθηκαν μόνο 57, ε, ε μόνο 57 αιτήσει ασύλου. Διαπιστώνουμε επίσης ότι κάποιε οργανώσεις αντιμετωπίζουν ε, δυσκολίες, όπως για παράδειγμα η Επιτροπή του Ελσίνκη, διότι το κράτος περιορίζει το περιθώριο ελιγμών τους ε, και το καθεστώς τους και ουσιαστικά η κυβέρνηση ε, πιέζει αυτές τις οργανώσεις για να μην δραστηριοποιούνται. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο ο Πρωθυπουργό μια χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ούγγρος Πρωθυπουργό, να αποκαλεί τους παράνομους μετανάστες εγκληματίες και λέει ότι η Ουγγαρία θα εφαρμόσει μια πολιτική που δεν θα επιτρέπει καθόλου μετανάστευση. Δήλωσε ότι η Ουγγαρία είναι πολιτιστικά ομογενής και δεν θα επιτρέψουμε να αλλάξει αυτό λόγω μετανάστευσης. Η ερώτηση μου λοιπόν προς τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τι σκοπεύουν να κάνουν ε, γι' αυτό, για το γεγονός δηλαδή ότι εφαρμόζεται μια τόσο περιοριστική πολιτική. Τι έχετε να απαντήσετε, τι επιλογές έχετε στη διάθεσή σας και πώς μπορείτε να πιέσετε προκειμένου να σταματήσει αυτή η πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πίτερ. Ο κύριος Κύρκος. Ευχαριστούμε για τη σημερινή σημαντική παρουσίαση. Οι εκθέσει αυτέ είναι σημαντικό εργαλείο για να διαπιστώνουμε τι αδυναμίε τη εφαρμογή τη νομοθεσία για το ζήτημα τη μετανάστευση και του ασύλου. Παρατηρούμε για άλλη μια φορά ότι οι χώρε στα σύνορα τη Ένωση δέχονται τι μεγαλύτερε πιέσει, το ξέρουμε και από τότε που γράφτηκε η έκθεση, οι πιέσει αυτέ γίνονται εκρηκτικέ. Γνωρίζουμε ότι η πρόσβαση στη διαδικασία του ασύλου δεν είναι πάντα εγγυημένη. Δεν μιλάμε για την αποδοχή ή όχι μια αίτηση, αλλά ούτε πρόσβαση. Και αυτή η πρόσβαση, η αδυναμία ε, προσέγγισης οδηγεί σε κινδύνους για τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό συμβαίνει κυρίως για αδυναμίες στην υπάρχουσα νομοθεσία. Η ευθύνη βέβαια πρέπει να πηγαίνει χέρι-χέρι με την αλληλεγγύη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενισχύσει τον καταμερισμό των ευθυνών μεταξύ όλων των κρατών των μελών, πιθανώς με ένα μηχανισμό που θα βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια. Είχαμε ένα ερώτημα για την αναφορά σας σε τρόπους ενίσχυσης των νόμιμων διάβλων μετανάστευσης. Υπάρχει έτοιμο κάποιο σχέδιο δράσης. Και τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στη Συμφωνία Επανεισδοχής με την Τουρκία. Το 2002 η Ελλάδα είχε υπογράψει με την Τουρκία μια αντίστοιχη συμφωνία διμερή η οποία οδήγησε σε 115.000 αιτήσει από την πλευρά της Ελλάδας και 4.000 απαντήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Τα νούμερα δείχνουν και το μέγεθος του προβλήματος. Η υπογραφή της νέας συμφωνίας του 2013 προσφέρει μεγαλύτερες εγγύησεις. Όμως, αφενός στη γειτονιά μας κάτι που αναβάλλεται για το μέλλον έχει τις περισσότερες πιθανότητες να μην υλοποιηθεί, αλλά και αφετέρου επειδή η κατάσταση στη γειτονιά της Ένωσης επιδεινώνεται διαρκώς και η πίεση θα είναι όλο και μεγαλύτερη, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια επιτάχυνση στην αντιμετώπιση του θέματος. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Μην αρχίσουμε τώρα όμως τους μακροσκελείς λόγους. Θέλουμε μια ελεύθερη σχετικά συζήτηση για το άσυλο, αλλά με βάση τα συγκεκριμένα θέματα. Παρακαλώ λοιπόν τους συναδέλφους να περιορίζονται στο λεπτό. Η κυρία Βεργία. με συγχωρείτε που το υπενθυμίζετε αυτό τη στιγμή που παίρνω εγώ το λόγο αλλά τέλος πάντων η παρουσίαση της έκθεσης αυτής είναι σημαντικό θέμα γιατί επαναφέρει την πραγματικότητα των αριθμών παρακαλώ κυρία Βεργία αν θέλετε παραπάνω από ένα λεπτό εντάξει γιατί και εγώ διαβάζω χωρίς τα γυαλιά μου και κάνουν πολλά λάθη, οπότε αν θέλετε παραπάνω από ένα λεπτό, σας παρακαλώ πέστε ό,τι θέλετε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να τα συμπυκνώσω. Τώρα έχασα ένα λεπτό όμως ήδη. Λοιπόν, έλεγα ότι αυτή η έκθεση ετήσια πάντοτε μας ξαναφέρνει στην πραγματικότητα των αριθμών. Καταρχήν θέτει την μετανάστευση προς την Ένωση στα πλαίσια της παγκόσμιας ε, μεταναστευτικών ροών και είναι σημαντικό και αυτό. Άλλο στοιχείο που επιτρέπει να σχετικοποιηθούν τα πράγματα είναι ότι η περισσότερη μετανάστευση αφορά τα πιο πολυπληθή κράτη-μέλη και αυτό πρέπει να τονιστεί και να σχετικοποιηθεί η σημασία του. Αν είναι σωστή αυτή η αριθμή τότε οι πέντε μεγαλύτερες χώρες της Ένωσης αντιπροσωπεύουν το 77% των μεταναστών. Όλοι ξέρουμε ότι η μεταναστευτική πίεση, όπως λένε, όρος που δεν μ' αρέσει, οφείλεται σε γεγονότα σε άλλες χώρες. Το 11 την Ίση έρχονταν στην Ένωση, σήμερα δεν ισχύει αυτό, σήμερα οι Σύριοι αποτελούν την κύρια μεταναστευτική ροή προς την Ένωση. Εξάλλου, με συγχωρείτε, αλλά και αυτό το μακάβριο παραλληλισμό που θα κάνω, βλέπετε και τον ρυθμό πνιγμένων στη Μεσόγειο. Σήμερα είναι Σομαλοί και Ερυθρέοι περισσότεροι. Πρέπει να το αναλύσουμε και αυτό σε σχέση με τα γεγονότα στις χώρες αυτές. Εχθές συνάντησα την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα αιτητών ασύλου και τρόμαξα από αυτά που μας είπαν για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι όσοι κρατούνται στα κέντρα μετανάστευσης οι περισσότεροι από αυτούς ζητούν άσυλο και κρατούνται μέχρι να διεκπαιρεωθεί η αίτησή τους και ακόμη πιο πολύ με τρόμαξα αυτό που μας είπαν για όσους έχουν ήδη το καθεστώς του πρόσφυγα την κατάσταση που αντιμετωπίζουν στην Ένωση. Αυτά που συμβαίνουν στην Ουγγαρία λοιπόν είναι σημαντικά και έχει πάρα πολύ μικρό αριθμό μεταναστών. Θα ήθελα να κάνουμε μια πραγματική αξιολόγηση του τι συμβαίνει για να μπορούμε να κάνουμε πραγματικές συγκρίσεις, να έχουμε συγκρίσιμα στοιχεία για την κατάσταση των μεταναστών στην Ένωση. Γιατί υπάρχουν τελείως απαράδεκτες καταστάσεις και για τους αιτητές ασύλου και για όσους έχουν ήδη τύχει μιας διεθνούς προστασίας. Γίνεται λόγος πολλής για τις συμφωνίες κινητικότητας και τις επιστροφές, αλλά δεν λέγονται και τόσο πολλά για την εθελοντική δίθεν επιλογή ορισμένων μεταναστών για να ενισχυθεί υποτίθεται η νόμιμη μετανάστευση. Να δούμε τι γίνεται ιδιαίτερα με την Τουρκία και την Τινησία. Γιατί και, στις δύο, και για τις δύο χώρες υπάρχουν συμφωνίες και επαναλαμβάνω ότι με ανησυχούν πολύ αυτά που γίνονται με τους Ερυθρέους διότι όλες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι σύλλογοι μας λένε ότι είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός τους που προσπαθεί να μπει στην Ευρώπη. Τελειώνω, τελειώνω κύριε Πρόεδρε. Δεν ενδιαφερόμαστε αρκετά λοιπόν για την κατάσταση στην Ερυθρέα. Είναι χώρα με την οποία σχεδόν ποτέ δεν έχουμε ασχοληθεί ενώ η κατάσταση εκεί είναι κρίσιμη λένε ότι είναι σαν ανοιχτή φυλακή, υπαίθρια φυλακή ολόκληρη η χώρα. Ξέρω πόσο ξεπέρασα το χρόνο μου, με συγχωρείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μάγερ. Μάγερ. Κυρία, κυρία Μάγερ, κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η πίεση στα εξωτερικά σύνορα αυξάνεται, ε, αυξάνονται οι αριθμοί και οι τραγωδίες στην θάλασσα. Η Κομισιόν συμφωνεί πως ε, ε, η πολιτική που ακολουθεί μέχρι στιγμής να φέρνουμε αυτούς τους ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τους ενθαρρύνουμε δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Thank you very much. I was, um, wrong footed by your brevity there. Ναι, με, με ευνηδιάσατε κιόλας, γιατί ήταν πολύ σύντομη η ερώτησή σας. Stevens, από το ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα είμαι σύντομη γιατί ε, είπαν αρκετά οι συνάδελφοι. Η κατάσταση των προσφύγων είναι δραματική και το αντιλαμβάνομαι πλήρως αλλά πρέπει να αντιληφθούμε πως και η Ευρώπη δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα όλου του πλανήτη. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Γι' αυτό έχω κάποιες ερωτήσεις προς την ε, Κομισιονίδα την έκθεση εγώ και θέλω να την ευχαριστήσω την Κομισιόν για την ενδιαφέρουσα αυτή η έκθεση. Αν δει κανείς λοιπόν το περιεχόμενό της, ο αριθμός των μπλε καρτών που δίνονται στην Ευρώπη για να προσελκύσουμε αποφύτους πανεπιστημίων ε, τους οποίους ε, χρειαζόμαστε ε, είναι μικρός, σχετικά μικρός θα έλεγα. Οπότε εγώ θα ήθελα να μάθω εάν η Κομισιόν σκοπεύει να κάνει κάτι για να αρθούν τα εμπόδια για ανθρώπους που είναι απόφτη πανεπιστημίων. Επίσης, διαβάζω αλλού στην έκθεση πως υπάρχει μια task force, μια ομάδα για τη Μεσόγειο και περιγράφονται διάφορα μέτρα. εγώ θα ήθελα να γνωρίζω σε ποιον βαθμό έχουν ληφθεί συγκεκριμένα αυτά τα μέτρα. Έχετε εφαρμόσει αυτό το σχέδιο. Έχετε κάποια αποτελέσματα. Και μια άλλη ερώτηση προς την Κομισιόν. Ε, η συμφωνία επανεισδοχής ε, που αναφέρατε με Τουρκία, Αρμενία και Πράσινο Κορτήριο είναι αυτές οι μόνες, ε, προετοιμάζεται και άλλες για να περιοριστεί ακριβώς το ποσοστό της μη νόμιμης μετανάστευσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τζιν Λάμπερτ. Uh, ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ και για την έκθεση. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον θέλει να σχολιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ποιες είναι οι τάσεις ε, για τα διάφορα ε, καθεστώτα προσφύγων και την επικουρική προστασία στα κράτη-μέλη. Όταν τα συζητήσαμε αυτά στην αναδιατύπωση της οδηγίας, είδαμε ότι κάποια κράτη-μέλη ε, εξέταζαν πολύ το θέμα της επικουρικής προστασίας, περισσότερο ως υποκατάστατο και όχι ως πρόσθετο της ανθρωπιστικής προστασίας. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον έχει κάτι να μας σχολιάσει από αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, υπάρχει μια έκθεση η οποία αναφέρεται στη χρήση κράτησης και το συνδέουν αυτό με πρόσβαση σε νομική συνδρομή και για το γεγονός ε, ότι πολύ συχνά είναι πολύ μικρότερη νομική συνδρομή για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται υποκράτηση. Και ίσως να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός των εφέσεων αν υπήρχε καλύτερη πρόσβαση σε νομική συνδρομή. Θα ήθελα τα σχόλιά σας επ' αυτού. Επίσης, υπάρχουν συστάσεις, ε, μας είπατε, στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και στις ε, εκθέσεις αναχώρα. Μπορείτε να μας πείτε λίγο καλύτερα το μηχανισμό γι' αυτό, γιατί πολλά από τα θέματα που συζητήθηκαν όσον αφορά την κοινωνική διάσταση είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει συνέπεια στην προσέγγιση που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Κάποια κράτη-μέλη ε, αναλαμβάνουν δράση για κάτι συγκεκριμένο και τους ζητάτε να αναλάβουν δράση, ενώ σε κάποιες άλλες χώρες στις οποίες δεν υπάρχει αντίστοιχη σύσταση παρά το γεγονός ότι υπάρχει αντίστοιχο πρόβλημα. Πώς θα προσεγγίζετε όλα αυτά. Και τέλος, ένας από τους άλλους τομείς ο οποίος μας ενδιαφέρει σε θέματα μετανάστευσης και συνδέεται λίγο και μετά όσα έλεγε και η κυρία Στίβενς, είναι το θέμα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων ε, των ε, υπηκών χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ συχνά ακούμε ότι η Στοκχόλμη έχει τους ε, καλύτερα καταρτισμένους ταξιτζίδες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει κάποια πρόοδος επ' αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Τζιν. Η κυρία Μπονιφή. Σε αυτή την ε, ανακοίνωση ε, διαπιστώνουμε ότι τα δικαιώματα των ετούντων άσυλο και των μεταναστών ε, ενισχύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεν, αλλά δεν φαίνεται ότι όπως μας είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, ότι είναι καλή διαχείριση όπως λέει η Ευρώπη φαίνεται ότι δεν έχει αντιληφθεί διδάγματα από το δράμα της ε, Λαμπεντούζας και σήμερα ε, προσπαθεί να έχει μια αποτελεσματική επιχείρηση για τη βοήθεια των μετανιστών και των ετούντων άσυλο που διασχίζουν τη Μεσόγειο για να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Είναι ανησυχητικά λοιπόν τα όσα γίνονται για την βοήθεια που προσφέρεται στους Σύρους πολίτες και επίσης ε, θεωρούμε ότι η βοήθεια αυτή είναι ανεπαρκής. Ε, είναι αρκετά τα μέτρα τα οποία υποτίθεται ότι ε, διεκδικούνται για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα ασύλου και παρόλα αυτά ο προπολογισμό για το άσυλο και τη μετανάστευση δεν αρκεί για να βοηθήσουμε και να έχουμε κατάλληλη φύλαξη στα εξωτερικά σύνορα. Πώ μπορούμε να έχουμε αποτελεσματικέ πολιτικέ όταν δεν υπάρχει κατάλληλο προπολογισμό. Πώ μπορούμε να βοηθήσουμε του ετούντε άσυλο και του μετανάστε όταν η πολιτική βούληση από πλευρά κρατών μελών είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η Ευρώπη θα πρέπει λοιπόν να είναι περισσότερο φιλόδοξη σε θέματα ασύλου και μετανάστευση. Θα πρέπει να ενισχύσει τον προπολογισμό τη ε, για τη βοήθεια των μεταναστών και των ετούντων άσυλο για να του βοηθήσει να ενταχθούν καλύτερα και η νόμιμη μετανάστευση θα πρέπει να γίνεται κατά προτεραιότητα σε συνεργασία με τις χώρες μετανάστευσης, μέσω συνεργασίας με τρίτες χώρες, όπως το επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να βοηθούμε και την ανάπτυξη αυτών των χωρών. Γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει πολύ περισσότερη φιλοδοξία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ. για την έκθεση. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και θα ήθελα να πω ότι επειδή αρχίζουμε να μπαίνουμε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης ε, λόγω της ε, κατάστασης στο Ιράκ ε, κατά του Ισλαμικού κράτους και επειδή ακριβώς δημιουργείται κατάσταση εκτάκτου ανάγκης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα κατεπηγόντως. Να σας αναφέρω μερικά αμοιβαία αναγνώριση καθεστώτος προσφύγων. Ήδη ακόμα δεν υπάρχει. Τι θέλουμε να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να το επιτύχουμε. Τι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να αντιμετωπίσουμε και την αδιαφορία πολλών κρατών μελών για την ε, ε, μεταφορά των προσφύγων. Στην σελίδα 7 της έκθεσης αναφέρεται ότι υπάρχει αδιαφορία και αυτό επιβεβαιώνεται και από τη στάση της Ουγγαρίας. Η εντολή της Frontex ακόμα δεν είναι ξεκάθαρη, δεν είναι σαφής ο ρόλος της και ποιος θα πληρώσει και το λογαριασμό. Οι νόμοι μεσοδοί για τη μετανάστευση δεν έχουν καμία εγγύηση. Αυτό σημαίνει ότι αφήνουμε ελεύθερο πεδίο στο οργανωμένο έγκλημα. Και Τέλος, διαφωνώ με την αισιοδοξία για την ε, μετεγκατάσταση των προσφύγων στην Ευρώπη. 15.000 πρόσφυγες μεταφέρθηκαν το 2013, αλλά υπήρχαν 300.000 αιτήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοράου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ρίξαμε μια ματιά στην ετήσια έκθεση για την κατάσταση ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013. Ακούσαμε και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από αυτά που μας είπε φαίνεται ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα σε σχέση με το παρελθόν. Εγώ εδώ είμαι πρωτόπυρος, δεν ξέρω πώς λειτουργούσαν τα πράγματα στο παρελθόν, αλλά βλέποντας τώρα τα πράγματα για πρώτη φορά διαπιστώνω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά το άσυλο στην Ευρώπη. Παραδείγματο χάρη, θα πρέπει να εξετάσουμε κατά την άποψή μου τους κανόνες ε, για το ποια είναι η χώρα που είναι αρμόδια για να λαμβάνει την αίτηση ασύλου. Το γεγονός ότι οι αιτήντες άσυλου θα πρέπει να βρίσκονται επί της ευρωπαϊκής επικράτειας. Ε, όσον αφορά το θέμα της αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, κατά την άποψή μου δεν είναι αρκετοί, ε, δεδομένου ότι υπάρχουν χώρε που λαμβάνουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων, όπω για παράδειγμα η Ιταλία. Και εκεί οι μεταναστευτικέ ροέ αυξήθηκαν κατά χιλιάδες ε, την τελευταία χρονιά και εξακολουθούν να αυξάνονται λόγω των ε, ε, πολέμων που είναι εξελίξει αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση, είναι σαφές ότι πρόκειται για εγκάρσιο ζήτημα, το οποίο δεν αφορά μόνο την Επιτροπή μας. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα εξωτερικής πολιτικής, το οποίο αφορά και τα όσα συμβαίνουν και στη Μεσόγειο. Το σύστημα της μπλε κάρτας φαίνεται ότι δεν ήταν ιδιαίτερα ε, αποτελεσματικό, διότι υπάρχουν ίσως κάποια κριτήρια τα οποία είναι πολύ αυστηρά και περιορίζουν πολύ τα πράγματα και ίσως θα έπρεπε να τα πλουστέψουμε λίγο περισσότερο για τους νόμιμους εργαζομένους. Τέλος, όσον αφορά το Frontex, Ακόμα θα θέλαμε να ξέρουμε ε, καλά ποια είναι τα ωριά της και ποια είναι η ακτίνα δράσης της υπηρεσίας αυτής και θα ήθελα να πω ότι όταν ε, ξεκίνησε στην Ιταλία η επιχείρηση Mare Nostrum, ε, άρχισε να συζητάτε το θέμα της διάθεσης στη θάλασσα, διότι θεωρώ με τη νέα ε, επιχείρηση θα είναι πολύ πιο δύσκολο να μπορέσει να διασώσει κάποιος στη θάλασσα ανθρώπους που έχουν βρεθεί εκεί. Ευχαριστώ. Θα κλείσω ο κατάλογος των ομιλητών. αν κάποιος θέλει να λάβει το λόγο, σας παρακαλώ να το δηλώσει τώρα. Αλλιώς κλείνει ο κατάλογος. Η κυρία ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάτι συγκεκριμένο για την επανεγκατάσταση. Η μόνη αναφορά που υπάρχει είναι στη σελίδα 7 με τέσσερις σιρούλες. Όλοι θυμόμαστε πέρσι πως ε, κάποιοι βουλευτές από τις νότιες χώρες είχαν ζητήσει μία συζήτηση για την επανεγκατάσταση μετά το πιλωτικό έργο που είχε ξεκινήσει στην Μάλτα. Η κυρία Μάλστρομ, η Επίτροπος, ήρθε και μας είπε ότι δεν θέλουν να το συζητήσουν καν τα κράτη-μέλη. Αναπάντεχο. Μετά από ε, μια τόσο σημαντική συνεδρίαση του Φόρουμ Επανεγκατάστασης θα έπρεπε να έχουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες, να ξέρουμε τι ε, σχεδιάζει η Κομισιόν για να συνεχιστούν αυτές οι συζητήσεις ε, για την επανεγκατάσταση γιατί για χώρες σαν τη Μάλτα η έννοια αυτή είναι κάτι το πολύ σημαντικό και προσφέρει μια λύση ή τουλάχιστον η συζήτηση ε, ελπίζουμε να οδηγήσει κάπου. Το μήνυμα που λαμβάνουμε είναι πως η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη δεν είναι διατεθειμένα να το συζητήσουν. Μόνο οι βουλευτές ε, σε συνεδριάσεις όπως αυτή εδώ ε, είναι διατεθειμένα να συζητήσουν. Αυτό δείχνει την αλληλεγγύη που υπάρχει. Ευχαριστώ. Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. η έκθεση αυτή, ε, ανάλογα με το ποιο τη διαβάζει, μπορεί να εξάγει διαφορετικά συμπεράσματα. Εγώ θα μπορούσα να σας πω ότι είναι χρήσιμη, ότι είναι απαραίτητη, ε, ότι είναι ανελιπής και ότι είναι τελείως συμβατική. Ανελιπής. Έχω 11 σημεία τουλάχιστον αξιολόγησης ε, για το άσυλο και τη μετανάστευση. Δεν θα ήθελα τώρα να, να κουράσω τους αδέλφους, διότι τα άκουσαν αρκετές φορές, αλλά υπάρχουν κάποια σχόλια τα οποία θα ήθελα να κάνω έτσι ενδεικτικά. Όπως ε, μόλις σας είπε και η Ρομπέρτα, το θέμα της επανεγκατάστασης ε, και όλα όσα έχουν σχέση με την κοινή αλληλεγγύη ε, κυρίως ε, όσον αφορά αυτές τις μικρές χώρες ε, που δέχονται τόσες πιέσεις σε θέματα ασύλου, δεν μπορεί να συζητάμε για την κοινή αλληλεγγύη με δυο γραμμές. Επίσης, δεν είμαστε σε θέση να έχουμε ένα νομοθετικό μέσο το οποίο να αναφέρεται σε κοινούς κανόνες αξιοπρέπειας. Στην οδηγία για τις επιστροφές ε, γίνεται αναφορά μόνο ε, στους χώρους κράτησης και τις προθεσμίες κράτησης, αλλά όχι για την αξιοπρέπεια και τις κατάλληλες συνθήκες κράτησης. Όσον αφορά τον κανονισμό Frontex, εκεί να σας πω ότι υπάρχει μια γενικευμένη σύγχυση. Μόλις άκουσα τον κύριο Κοράο, τον οποίο σέβομαι ιδιαίτερα και μόλις ήρθε, αλλά ε, να σας πω ότι ο Frontex δεν είναι υπηρεσία ε, θαλάσσιας διάσωσης. Ευτυχώς όμως διασώζει ανθρώπους στη θάλασσα, ε, διότι η Frontex είναι συνεργασία, αλλά η Frontex είναι και μια υπέροχη ιδέα μεν που δεν έχει εφαρμοστεί καταλήλως. Υπάρχει το CRADE που είναι ένας κατάλογος ε, προσφοράων ε, που δεν ε, υλοποιήθηκαν ποτέ. Ο Frontex δρά μόνο όταν τον φωνάζουν. Πρέπει κάποιος να φωνάξει για να έρθει η ευθύνη του ελέγχου των συνόρων είναι ευθύνη της κάθε χώρας και ο Frontex ε, ε, είναι θέμα συνεργασίας. Θα πρέπει όμως να αναφερθούμε και στην ε, μοναδικότητα και των αέριων συνόρων και των χερσαίων συνόρων. Όπως υπενθύμησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι εθνική αρμοδιότητα κάποια θέματα, είναι σαφής επικουρικότητα. Επομένως θα πρέπει να γίνουν συστάσεις και στο θέμα αυτό αλλά και σε άλλους τομείς. Αλλά θα ήθελα να ξέρω και δύο λόγια για την χρηματοδότηση του νομοθετικού μέσου για τα FEE e σύνορα. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε συζητήσει, αλλά είναι αρκετά περίπλοκο. Ένα δις ε, εκατό εκατομμύρια για να ξεκινήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και λίγο το δόγμα των Ηνωμένων Εθνών σε θέματα μετανάστευσης και ανάπτυξης. Ε, πολλές φορές ε, οι επιστροφές για τα κράτη-μέλη είναι πολύ σημαντικό τμήμα του ΑΕΠ τους και του πλούτου τους. Και ολοκληρώνοντας θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να δούμε λίγο και τις συστάσεις και την επικουρικότητα και το κατά πόσο θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί ποινικοί κώδικες για να τιμωρούνται πολύ αυστηρά οι έμποροι, οι άνθρωποι οι οποίοι παίζουν με την επιπλησία των ανθρώπων. Και τέλος, κύριε Πρόεδρε, να σας πω για άλλη μια φορά, όπως ε, γνωρίζετε ο, ο συνάδελφος, ο προηγούμενος πρόεδρος Χουάν Χορνάντος ε, Λόπες Αγγιλάρ, δεν θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε ποτέ τον όρο παράνομος. Αναφερόμαστε σε παράτυπους, ε, αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος παράνομος σε καμία περίπτωση. Αυτά δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Thank you, Mr. Diaz for the, the last point. It's uh, also a good reminder also for our new members about um, Ευχαριστούμε κύριε Μέρες. Πολύ καλή υπενθύμηση και των διαδικασιών και της ορολογίας που χρησιμοποιούμε. Τέλος, έχουμε δύο ακόμα ομιλητές, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, η κυρία Γουίμπεργκ Ευχαριστώ. Εγώ κατάγομαι από μια χώρα, τη Σουηδία, που είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που έχει ε, από τις περισσότερες αιτήσει ασύλου και μεταναστών. Και φυσικά είναι πολύ μεγάλο το κόστος από αυτές τις δραστηριότητε και δεν έχουμε τη δυνατότητα να υποδεχόμαστε με αξιοπρέπεια αυτούς τους ανθρώπους. Θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες προποθέσει, να υπάρχουν και κάποιοι ε, χώροι υποδοχής των μεταναστών και ε, φαίνεται ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται επί τόπου ε, ε, αναφέρεστε φυσικά στα όσα συμβαίνουν, ξέρουμε και τι γίνεται και στη Συρία, πρέπει να το βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς, αλλά θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται, να δούμε πώς γίνονται τα πράγματα, θα πρέπει να έρθει και κάποιος επιτόπου και για να φτάσει κάποιος σε εμά έχει διασχίσει πάρα πολλές χώρες. Ε, είναι δυνατόν να μην ελέγχεται ποιο περνάει από τα σύνορα, ε, πρέπει να ελέγχονται κάπως αυτές οι ροές μεταναστών. Θα πρέπει λοιπόν να, δω και, να δούμε και τι γίνεται και να δούμε και τι γίνεται στα σύνορα, διότι ορισμένες φορές αναγκαζόμαστε εμεί να πληρώνουμε το τίμημα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν πολύ συγκεκριμένοι. Τελευταίος ο μιλητής, ο κύριος ε, Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Εδώ δεν βλέπω προοπτικές στην έκθεση αυτή. Απλά διαπιστώνουμε πως ο αριθμό των ετούντων άσυλο αυξάνεται, το ξέρουμε αυτό. Αλλά ο Ματέο Ρέντσι ήρθε στην επιτροπή μας, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, κύριε πρόεδρε, και μας είπε πως προσεχώς δεν πρέπει να κάνουμε τους παράνομους νόμιμους, αλλά θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις αιτίες. Ε, ειδικά να μιλάμε για φτωχούς ε, και τα λοιπά. Να βρεθεί ένας τρόπος να αποκτήσουν προοπτική. Τι σκέφτεστε, γιατί δεν υπάρχει τίποτα σε αυτή την έκθεση. Επίσης για τα λόμπι επίσης των λαθρεμπόρων που υπάρχουν και δραστηριοποιούνται. Τι σκοπεύετε να κάνετε εναντίον αυτών. Επίσης, ε, το σύστημα της ε, μπλε κάρτας από ό,τι φαίνεται μόνο στη Γερμανία εφαρμόζεται. Στις υπόλοιπες χώρες όχι. Σας ευχαριστώ. Είναι χρήσιμη νομίζω η συζήτηση παρά το ότι έπρεπε να έχουμε διαβάσει την εκθεσή ούτως ή άλλως να δούμε το που τοποθετούνται και οι βουλευτές ε, στα ευρύτερο αυτό ζήτημα πριν περάσουμε στους συγκεκριμένους φακέλους. να ακούσουμε και τις δύο πλευρές. Ήταν χρήσιμη λοιπόν νομίζω η συζήτηση. Τώρα να προσθέσω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Διαβάζοντας ε, την ε, έκθεση δεν υπάρχει τίποτα για την εφαρμογή. Η ανησυχία που έχουμε είναι πως ε, αυτό το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε έχει γίνει. Δηλαδή ήταν νομοθετικό το έργο, ειδικά όσον αφορά το πακέτο του ασύλου, το ζήτημα είναι η εφαρμογή. Και η έκθεση εδώ πέρα γράφει το τι δεν κάνουν τα κράτη-μέλη, συλλογικά ή μεμονωμένα, δεν εφαρμόζεται η οδηγία κτλ. Έχετε να μας πείτε κάτι από αυτού. Και τέλος για την νόμιμη μετανάστευση ε, τους ε, εποχικούς ε, εργαζόμενους βλέπουμε πάλι το μέλλον της εφαρμογής σε ένα εχθρικό πολιτικό κλίμα και ε, η κυρία Σίπολ ανέφερε το μέλλον των υπολείπων πτυχών ε, της ε, νόμιμης μετανάστευσης, φοιτητές, επισκέπτες κτλ. Με τα υπόλοιπα ζητήματα τι γίνεται. Σε ένα αρκετά εχθρικό θα έλεγα πολιτικό κλίμα για την νόμιμη μετανάστευση. Έχετε τον λόγο και ο κύριος Ράιν νομίζω έχει να πει κάποια πράγματα για το άσυλο. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις. Θα αναφερθώ στα βασικά της μετανάστευσης και για το άσυλο θα δώσω τον λόγο συνάδελφο. Από την τελευταία ερώτηση να ξεκινήσω για την εφαρμογή και το μέλλον. Οπωσδήποτε είναι προτεραιότητα για την επόμενη Κομισιόν. Νομίζω αυτό αναφέρθηκε ήδη από τον Πρόεδρο και όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση. Υπάρχει ένα επαρκές ε, σώμα νομοθεσίας που έχει ε, ήδη εγκριθεί. Έχουμε 8 τομεακές οδηγίες και μία ακόμη υποδιαπραγμάτευση. Οπωσδήποτε η εφαρμογή λοιπόν θα είναι προτεραιότητα όπως και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ε, των οδηγιών αυτών. Όσον αφορά τη μετανάστευση έχουμε κάποιες μελέτες ε, που συνεχίζονται και αφορούν βέβαια και τον αντίκτυπο και τα δικαιώματα των ε, υπηκών τρίτων χωρών. Όσον αφορά οπωσδήποτε το μέλλον, ο Επίτροπος την επόμενη εβδομάδα θα τα αναπτύξει στις ακροάσεις, ε, ο υποψήφιος Επίτροπος, αλλά μπορώ να σας ε, πω πως ε, στις προγραμματικές δηλώσεις του Πρόεδρου Γιούνκερ αφορά... Ε, περιέχονται πολλά πράγματα για την μπλε κάρτα και τους ανθρώπους υψηλής εξειδίκευσης και τονίζει το ότι έχουμε ένα, δύο το πολύ κράτη-μέλη που εκδίδουν τις περισσότερες μπλε κάρτες, ενώ δεν έχει επιτύχει το σύστημα αυτό στα άλλα κράτη-μέλη. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν την εξέταση αυτού του ζητήματος και η πρώτη έκθεση εφαρμογής της μπλε κάρτας ε, ε, εκδόθηκε τον Μάιο. Είχα μια πρώτη ανάλυση με βάση τα εφιστάμενα δεδομένα. Προωθούμε την ανάλυση μας και στους επόμενους μήνες θα έχουμε την ε, εξέταση της εφαρμογής για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση, για να γίνει πιο ελκυστική η Ευρωπαϊκή Ένωση για ανθρώπους ε, υψηλών ικανοτήτων και να δούμε τι αλλαγές ε, χρειάζονται. Επίσης, αυτό το οποίο τονίζουμε είναι πως οπωσδήποτε το ότι υπάρχουν εθνικά συστήματα τα οποία επιτρέπει η οδηγία για ανθρώπους με υψηλές δεξιότητες ε, δεν δημιουργεί ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο. Οπότε τα κράτη-μέλη βγάζουν κάποιες άδειες ε, για ανθρώπους με ικανότητες, αλλά οπωσδήποτε ε, δεν είναι μπλε κάρτες, οπότε δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και ποιοι είναι οι κανόνες για να προσελκύουμε τέτοια άτομα. Θα το δούμε λοιπόν αυτό πάρα πολύ προσεκτικά στο μέλλον. Επίσης, ετέθη το ζήτημα του πώς θα γνωστοποιήσουμε τις νόμιμες διόδους ε, μετανάστευσης. Υπάρχει ένα πόρταλ. Υπάρχουν πληροφορίες για τις οδηγίες ε, και για τις εθνικές διαδικασίες ε, και συνδέσμους. Βεβαίως δεν αρκεί αυτό και σκοπεύουμε να το αναβαθμίσουμε αυτό, να υπάρξει μεγαλύτερη διάδοση και ένα άλλο κομμάτι θα είναι οι εκστρατείες ενημέρωση θα κάνουμε σε τρίτες χώρες, ειδικά στην Αφρική και θα καλύψουν και τη δυνατότητα των νόμιμων διόδων. Επίσης, υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις ε, για το οργανωμένο έγκλημα και την ε, ελαφρέα είσοδο μεταναστών, ειδικά κάτι το οποίο αφορούσε την ε, ομάδα εργασίας ε, για την ε, Μεσόγειο. Συνεργαζόμαστε με διάφορους ενδιαφερόμενους να δούμε το τι γίνεται, όπως είπα, για την δίωδο αυτή με την Frontex και τη Europol συνεργαζόμαστε και την ε, ΕΑΖΟ, την υπηρεσία του ασύλου, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο που είναι πράγματι μία από τις αιτίε. Και θα καταρτήσουμε αρχές του επομένου έτους ένα σχέδιο δράσης για να κάνουμε κάτι και βεβαίως μιλάω και για επιχειρήσεις, επιχειρησιακές δραστηριότητες, συνεργασία μεταξύ της ε, Europol και της Frontex και των κρατών μελών ιδιαίτερα. Η καταπολέμηση λοιπόν του οργανωμένου εγκλήματος ε, και των ε, δουλεμπόρων είναι ένα από τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Επίσης υπήρχαν πολλά ερωτήματα που αφορούσαν τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης. Όπως τονίσαμε και στην ανακοίνωσή μας στην ομάδα εργασίας για τη Μεσόγειο, είναι βασική αυτή η πτυχή. Πρέπει να συνεργαστούμε με τις τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης και έχουμε ε, ήδη διαδικασίες ε, συζήτησης και συνεργασίες με τις χώρες αυτές. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Ο πολιτικός διάλογος ε, με τις χώρες στο κέρας της Αφρικής, η λεγόμενη διαδικασία του Χαρτούμ, θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο ε, ήδη δηλαδή, ξεκινήσει η πολιτική ας πούμε έναρξη θα γίνει το Νοέμβριο, θα συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές στο κέρας της Αφρικής για να ενισχυθεί η διαχείριση λιμένων και κοινή καταπολέμηση λαθρεμπορίου εμπορευμάτων και διακίνηση ανθρώπων. Επίσης ανέφερα την ε, συμφωνία κινητικότητας με την Ισία και Μαρόκο. Αυτό δεν αφορά μόνο τις επανεισδοχές, ε, και αυτό αφορά βεβαίως, αλλά είναι επίσης κάτι το οποίο αφορά ε, πρώτα απ' όλα και την πληροφόρηση για εκπαίδευση, νόμιμες διόδους ε, και εκπαίδευση για επικοστρίτων τρίτων χωρών που θα εργαστούν σε κάποιο κράτος μέλος. Προσπαθούμε λοιπόν να προωθήσουμε μια συνολική προσέγγιση όσον αφορά την ε, ε, συμφωνία αυτή και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και την ενίσχυση της νόμιμης. Υπήρξαν επίσης κάποιες ερωτήσεις ε, για τους συνοριακούς ελέγχους και τον ρόλο της Frontex. Η Κομισιόν, όπως έχει επισημάνει και η κυρία Μάλμστρομ και ο κύριε Γενικός μας Διευθυντής, ε, η Frontex δεν είναι ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή. Είναι ένα, μια επιχειρησιακή υπηρεσία η οποία συντονίζει τις δραστηριότητες των κρατών μελών όσον αφορά την επιτήρηση και τον έλεγχο των συνόρων. Βεβαίως ε, προτεραιότητα δίνουν στα εξωτερικά εκείνα σύνορα όπως τη Μεσόγειο όπου υπάρχει ανάγκη και έτοιμα από τα κράτη-μέλη. Αλλά δεν έχει δίκου της πόρους, ε, βασίζεται η Frontex ε, στη συνεργασία των κρατών μελών. Όλων των κρατών μελών. Γι' αυτό η Κομισιόν πάντα ζητούσε περισσότερες συνεισφορές ε, από τα άλλα κράτη-μέλη στις κοινέ επιχειρήσεις που συντονίζονται και υποπτεύονται από τη Frontex και ειδικά για να στηριχθούν οι δράσεις στη Μεσόγειο. Τώρα οι συζητήσεις ε, συνεχίζονται με τη Frontex και τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη για το πόσο μπορεί να αναβαθμιστεί το έργο της, ειδικά στη Μεσόγειο, με την επιχείρηση τρίτων, νομίζω θα λέγεται, η οποία δεν θα αντικαταστήσει τη Mare Nostrum, αλλά θα αυξήσει την παρουσία της Frontex και τις ε, κοινέ επιχειρήσεις των κρατών μελών στη Μεσόγειο για να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη που είναι πιο εκτεθειμένα. Νομίζω. Α, ναι, για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ναι. Υπήρχε μία ερώτηση σχετικά. Όπως ξέρετε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Οπωσδήποτε αφορά κυρίως οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές. Αλλά φέτος συνεργαστήκαμε στενά με τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και άλλες γενικές διευθύνσεις για να διασφαλίσουμε πως θα έχουμε συγκεκριμένες συστάσεις ε, όπου, για τις χώρες εκείνες όπου υπάρχει μεγάλο κενό ας πούμε στο ποσοστό απασχόλησης ε, ε, μεταναστών σε σχέση με τους υπηκόους π.χ. Βέλγιο, Σουηδία όπου υπήρχε ακριβώ αυτό το κενό με τους υπηκόους τρίτων χωρών Προσπαθούμε δηλαδή να ενεργοποιηθεί στην αγορά εργασίας ο πληθυσμός των μεταναστών και άλλα μέτρα κοινωνικής ε, ε, ένταξης και να υπάρχουν περισσότερες ε, συνέργειες μεταξύ μετανάστευσης αφενός και οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών αφετέρου. Θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η διαδικασία και θα την ενισχύσουμε. Νομίζω πως οι περισσότερες ερωτήσεις απαντήθηκαν. Θα δώσω λόγο στον Στίβεν για να σας πει τα του ασύλου και της ε, διεθνούς προστασίας. Thank you, Lara. Ευχαριστώ, Λάρα. Ναι, σύντομα, ε, σύντομα, ορίστε. Ναι, θα είμαι συντομότατος. Πρώτον, εισαγωγικά. In the area, the focus... Για το άσυλο, εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι τα επόμενα χρόνια η βάση θα είναι η εφαρμογή, όπως είπε και ο κύριος Μωράης και ο Λάρη, η Λάρα. Έχουμε τώρα ένα σαφές νομικό πλαίσιο και πολλά από τα ερωτήματα που τέθηκαν δείχνουν ότι η μεγάλη πρόκληση θα είναι πώς θα τα εφαρμόσουμε όλα αυτά στην πράξη. Όχι μόνο για να βοηθηθούν οι χώρες μέλη, αλλά και για να έχουμε περισσότερη γνώση για το τι συμβαίνει σε ολόκληρη την Ένωση, σε όλα τα κράτη-μέλη, με τη βοήθεια βέβαια της υπηρεσία μας στη Μάσχα, στη Μάλτα, με συγχωρείτε. Τώρα, για τα συγκεκριμένα από δουλευτάς Ένας ρώτησε για την κατάσταση στην Ουγγαρία. Η Κομισιόν γνωρίζει ότι υπάρχουν προβλήματα στην Ουγγαρία με την εισρωή περισσότερων αιτητών ασύλου και μεταναστών. Και αυτό είναι πρόσφατο και δημιουργήθηκε τεράστιο πρόβλημα για την υποδοχή τους. Ήρθαμε σε επαφή με τις Ουγγαρικές αρχές, επισκεφτήκαμε κέντρα εκεί και διαπιστώσαμε σημαντικές βελτιώσεις αν και δεν είναι ακόμη ιδεώδη τα πράγματα. Υπήρξαν όμως σημαντικές βελτιώσεις παρομοίως. Ο Ούγκρος βουλευτής ανέφερε τις ανησυχίες που έθεσε η Επιτροπή Ελσίνκη Ουγγαρίας. και τις ανησυχίες αυτές τις θέσαμε και εμείς στις Ουγγρικές Αρχές, ιδίως για τις συνθήκες κράτησης. Και εκεί σημειώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις που πρέπει να τις αναφέρουμε. Δεν πρέπει να τις αγνοήσουμε, αλλά παραμένουν ακόμη ορισμένα προβλήματα που ακόμη τα συζητούμε με τους Ούγγρους. Τώρα τα υπόλοιπα ερωτήματα που τέθηκαν. Versia asked κυρία Βέρζιο ρώτησε κάτι για τη χρήση της κράτησης και τις συνθήκες στα κέντρα κράτησης. Υπάρχει, επαναλαμβάνω τώρα, ένα ρητό σαφές νομικό πλαίσιο που δείχνει ότι η κράτηση των ε, αιτητών ασύλου πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε επίγουσες και ακραίες καταστάσεις και διασαφίζει ότι η κράτηση πρέπει να εφαρμόζει ορισμένα κριτήρια και πρότυπα και θέλουμε αυτό να εφαρμοστεί και να γίνει σεβαστό σε όλες τις χώρες μέλη. Η κυρία Μάγερ, η Μα Λάμπερτ, ρώτησε για τη χρήση των, από χώρες μέλη των διαφόρων καθεστώτων αναγνώρισης του πρόσφυγα, του καθεστώτος του πρόσφυγα ή της συνοδευτικής προστασίας. Θα ήθελα απλώ να πω ότι το νομικό πλαίσιο είναι σαφές, για τρίτη φορά το λέω, και ότι είναι σαφή τα κριτήρια για το ποιος μπορεί να θεωρηθεί επισήμως ως πρόσφυγας. Ξέρουμε ότι στην πράξη υπάρχουν ακόμη διαφορές στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν το νομικό αυτό Υπήρξε όμως κάποια σύγκληση και είναι από τα θέματα που συνεχίζουμε να εξετάζουμε και αυτό ισχύει και για την υπηρεσία της Μάλτας. Με τα κράτη-μέλη κάνουμε μια διαπαιδαγωγική δραστηριότητα αυτή τη στιγμή για να δούμε πώς ακριβώς πρέπει να εφαρμόζονται όλα αυτά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ελπίζουμε με τον καιρό να υπάρξει σύγκληση στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται ή χορηγούνται αυτά τα καθεστώτα. Επίσης πολλά ερωτήματα τέθηκαν για την αλληλεγγύη γενικότερα. και τέθηκαν συγκεκριμένες ανησυχίες, εκφράστηκαν από τον βουλευτή από την Μάλτα για την εγκατάσταση ορισμένων προσφύγων από δική μας πλευράς και αυτό το είπε επανειλημμένος ο πρώην Επίτροπος και είμαι βέβαιος ότι θα το συνεχίσει και ο επόμενος οι πρακτικές εγκατάστασης relocation είναι βασικό στοιχείο της αλληλεγγύης και φαντάζομαι ότι τα κράτη-μέλη θα τη χρησιμοποιούν πολύ σπάνια. Η Μάλτα έχει ωφεληθεί από αυτή την πρακτική μέχρι σήμερα αλλά στο μέλλον μπορεί να υπάρξουν καταστάσεις όπου οι χώρες, μερικές χώρες, θα πρέπει να έχουν αρκετή πολιτική θέληση για να μεταφέρουν αλλού τους μετανάστες εφόσον έχουν σημαντικό πρόβλημα απορρόφησης του αριθμού των μεταναστών ή προσφύγων. Αλλά παραμένει εθελοντική, προαιρετική. Παρακαλώ να καταλήγεις, Σίβεν. Ναι, καταλήγω με το εξής. Έχουμε δώσει οικονομικά κίνητρα στα κράτη-μέλη και το ετήσιο forum relocation που αναφέρατε προηγουμένως θα ξανασυνεδριάσει το Νοέμβριο φέτος και θα το χρησιμοποιήσουμε σαν μια ευκαιρία για να ζητήσουμε πάλι από τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν την πρακτική αυτή όποτε και όπως πρέπει. Τώρα επειδή λείπει ο χρόνος ας σταματήσω εδώ νομίζω όμως ότι κάλυψα τα κύρια ερατήματα. Νομίζω ότι τα καλύψατε και οι δύο και συγγνώμη που σας διακόπτω γιατί θα μπορούσαμε να το συζητάμε ώρες. Ε, οι επικρίσεις είναι πολύ σημαντικές, είναι πολύ σημαντικό για μας. Ε, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που βασικά αναφέρθηκαν στις βασικές πτυχές γιατί έχουν μεγάλη σημασία ε, γιατί είναι καλό να σταθούμε στην ουσία της έκθεσης και θα πρέπει να απαντήσουμε και επισήμω στην έκθεση αυτή. Ε, θεωρώ ότι ήταν χρήσιμη λοιπόν η συζήτηση. Μπορούμε να έχουμε τώρα μια συζήτηση η οποία θα επικεντρωθεί καλύτερα ε, στο, ε, στην ΕΑΣΟ, στην Υπηρεσία Σύλλου. ξέρετε όμως ότι βρισκόμαστε και σε μια κρίσιμη στιγμή σε αυτή τη συζήτηση γιατί συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μεσόγειο και είναι κατάλληλη στιγμή λοιπόν για να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι και η Τζιν Λάμπερτ εδώ, η οποία είναι η για την ΕΑΣΟ, καθώς επίσης και συνάδελφοι που είναι εισηγητές ε, για θέματα ασύλου, το οποίο συζητήσαμε και στην προηγούμενη συζήτηση. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα είναι ιδιαίτερα επικοδομητική συζήτηση και για τα μέλη ε, που ε, είναι καινούρια το θέμα του ασύλου δεν συζητάται μόνο από την πλευρά της υπηρεσίας του ασύλου ως υπηρεσία, αλλά κοιτάμε να δούμε και τι δεν λειτουργεί. Ακούγεται συνέχεια όρος αλληλεγγύη, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας και βεβαίως ε, η έκθεση θα παρουσιαστεί. Μας είπατε ότι θα κάνετε μια σύντομη ε, δήλωση και μετά θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις και στη συνέχεια θα επανέλθετε. Αντί να ακούσουμε λοιπόν μια μακρισκελή δήλωση, ε, θα ε, συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Υπάρχει και το πολιτές πρόγραμμα εργασίας. Καλό θα ήταν λοιπόν να σταθείτε στις βασικές πτυχές και από εκεί και πέρα να δούμε τι ερωτήσεις υπάρχουν και να επανέλθετε, να είναι λίγο πιο ευέλικτος ο ο τρόπος που θα συζητήσουμε. Να, βασι... να αναφερθείτε στα βασικά στοιχεία και από εκεί και πέρα να δούμε τι ε, θα προκύψει από τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και θα θέλαμε να ακούσουμε τα σχόλιά σας. Αξιότιμα κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ καταρχάς για τη νέα κοινοβουλευτική θητεία και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και την κατάλληλη έμπνευση για τη δουλειά σας. Μπορείτε σίγουρα να βασιστείτε στην πλήρη υποστήριξή μου ε, και στην πλήρη υποστήριξη από πλευρά της υπηρεσίας μας. Θα είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομος για να ε, διευκολύνω τη συζήτηση. Για να διευκολύνω τη συζήτηση σας έχει διανεμηθεί, ελπίζω να το λάβατε, και ένα σύντομο έγγραφο το οποίο συνοψίζει τις βασικές εξελίξεις αυτή τη στιγμή. Ο βασικός λόγος ε, για τον οποίο βρίσκομαι εδώ είναι η ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ασύλου και ήδη προς μεγάλη μου χαρά έχει γίνει έγγραφο το οποίο χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς και ελπίζω να χρησιμοποιηθεί αυτό και στο μέλλον, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε έτσι και να αποτελεί ένα πρακτικό οδηγό για την κατάσταση του ασύλου. Αν δούμε τι συνέβη την προηγούμενη χρονιά, γιατί κυρίως η έκθεση αναφέρεται στην προηγούμενη χρονιά, Υπάρχουν τρεις βασικές ροές ε, το 2013. Η Συρία, η Ρωσική Ομοσπονδία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Αν εξετάσουμε τις διάφορες ροές, βλέπουμε τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Για τη Συρία νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας πω λεπτομέρειες. Η κατάσταση είναι γνωστή, τη βλέπετε καθημερινά στις οθόνες της τηλεόρασής σας και ήδη ε, από τον τελευταίο μήνα έχουμε όλο ένα και αυξανόμενους αριθμούς οι αιτήσει σύρων πολιτών ε, βρίσκονται μεταξύ των πρώτων τριών αιτήσεων ασύλων ε, μεταξύ 19 κρατών μελών. Αυτό ε, δείχνει πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Η Ρωσία είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Πέρσι είχαμε μια σημαντική αύξηση, αλλά προς το τέλος του έτους μειώθηκε ουσιαστικά. Αν δούμε και το είδος των αιτήσεων, διαπιστώνουμε ότι οι αιτήσει από τη Ρωσία μπορεί να είναι από Τσετσένους και κυρίως αυτές ε, απορρίπτονται στην πλειονότητά τους. Στα Δυτικά Βαλκάνια είναι τελείως διαφορετικά τα χαρακτηριστικά επίσης. Στα Δυτικά Βαλκάνια έχουμε μια κατάσταση η οποία διονύζεται εδώ και αρκετά χρόνια και το ίδιο είχαμε και στο πρώτο εξάμεινο του έτους και είναι πολύ σημαντικό τμήμα των μεταναστευτικών ροών και έχουμε ε, πολλές απορρίψεις. Το ποσοστό απορρίψης είναι περίπου 96% και σε κάποιες περιπτώσεις ε, φτάνει και στο 100%. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Οι Σύριοι λοιπόν την χάνουν προστασίας, δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω τους λόγους και τα άτομα από τα Δυτικά Βαλκάνια συνήθως δεν θεωρούνται άτομα τα οποία πρέπει να ε, έχουν προστασία. Οι πιο πρόσφατες εξελίξεις τώρα και τάσεις για το πρώτο εξάμεινο του φετινού έτους ε, διαπιστώνουμε ότι οι τάσεις που είχαμε πέρσι, ε, ε, διότι πέρσι είχαμε τον υψηλότερο αριθμό από τότε που άρχισε να συλλέγει στοιχεία η Eurostat, εξακολουθούν να αυξάνονται. Αναφέρθηκα στη Συρία, έχουμε το Ιράκ και την Ουκρανία στη συνέχεια και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι και τους λόγους. Η Ερυθρέα ξεπετάχτηκε και αυτή στην εικόνα ξαφνικά. Ε, μέχρι τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς γιατί. Η κατάσταση στην Ερυθρέα ήταν πολύ κακή εδώ και πολλά χρόνια. Ξακολουθεί να είναι πάρα πολύ κακή, αλλά αυτό από μόνο τους δεν εξηγεί αυτή την ξαφνική αύξηση. Ε, Το εξετάζουμε με τα κράτη-μέλη και εμπειρογνώμονες για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Τώρα, αυτό το οποίο κάναμε πέρσι και φέτος ε, κυρίως ήταν να επικεντρωθούμε ε, στη βοήθεια προς τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή του κεκτημένου όσον αφορά το άσυλο. Ε, πέρσι έγινε δεκτή η πρόταση για το η δέσμη μέτρων για το άσυλο, πολύ σημαντικό βήμα και από εδώ και πέρα έχουμε περάσει στην εφαρμογή και όλοι πρέπει να εφαρμόσουν αυτά τα οποία υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν. Αυτό γίνεται με κοινά προγράμματα κατάρτισης, με εκπόνηση εγχειριδίων τα οποία θα μας επιτρέψουν να εφαρμόσουμε με πρακτικό τρόπο την νομοθεσία που εγκρίθηκε να υπάρχουν πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής. Ε, πέρσι έγινε μια μελέτη για την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια. Όπως ε, σας είπα, η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες ε, για τους οποίους υπάρχουν πιέσεις αλλά και επιστροφές στα Δυτικά Βαλκάνια. Και πολύ σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα στι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μία έκθεση για την Τσετσενία και σε μερικέ εβδομάδε θα έχουμε και μία έκθεση για τη Σομαλία και ετοιμάζουμε και μία επικαιροποίηση της κατάστασης ασφαλείας ε, στο Αφγανιστάν. Ε, εξετάζουμε λοιπόν διάφορες χώρες καταγωγής και ε, ταυτόχρονα προσπαθούμε να έχουμε και κάποιους εμπειρογνώμονες για το Ιράκ, τη Συρία, την Ουκρανία και άλλες περιοχές οι οποίες είναι σημαντικές αυτή τη στιγμή. Αναφέρθηκα κύριε Πρόεδρε και ε, επειδή θα θέλω να τηρήσω το λόγο μου και να είμαι σύντομος, ε, όσον αφορά τα σχέδια για τη Μεσόγειο, εκεί είχαμε μια αναφορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν χρειάζεται να σας πω εγώ πολλές λεπτομέρειες, δύο πράγματα ίσως. Πρώτον, έχουμε ξεκινήσει επιτέλους να πω, διότι ήταν ένα θέμα το οποίο ήδη από το πρόγραμμα της Χάγης του 2004 ε, σημαντικό. Έχουμε αρχίσει λοιπόν κάποια πρώτα βήματα για την ε, διαδικασία της κοινή επεξεργασίας και είναι τα πρώτα δειλά βήματα τα οποία είναι ιδιαίτερα εθαρρυντικά. Δεύτερον, συνεργαζόμαστε με τη Europol, τη Frontex και τη Eurojust, ε, ένας πολύ ενδιαφέρον συνδυασμός, για ένα πρόγραμμα στη Μάλτα και ένα πρόγραμμα στην Ιταλία, προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη εικόνα του φαινομένου των εγκληματικών οργανώσεων που ε, βρίσκονται πίσω από τις μεταναστευτικές ροές. Ένας πολύ σημαντικός και νέος τομέας ε, και φαντάζομαι ότι θα επανέλθουμε εν ευθέτω χρόνο σε αυτό. Φυσικά μπορούμε να εργαστούμε όταν έχουμε κατάλληλο προπολογισμό και ανθρωπίνου πόρου. Και γι' αυτό ακριβώ θα ήθελα να, βοηθήσω την, να ευχαριστήσω την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για την τροπολογία τη. Σα ευχαριστώ θερμά, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, αναγνωρίζει το γεγονός ότι χωρίς ε, κατάλληλους ανθρώπους δεν μπορούμε να εργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Ρόμπερτ και σε ευχαριστώ που ήσουν και σύντομο, διότι έτσι μπορούμε να συζητήσουμε και να επανέλθει στη συνέχεια ε, μετά τα σχόλια. Συνάδελφοι, ε, προφανώς υπάρχει το επιχειρησιακό σκέλος ε, του τι κάνει το ΙΑΣΟ και θα ήθελα να επικεντρωθείτε σε αυτό, αλλά υπάρχει και το θέμα της ποιότητας του ασύλου και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και τα πολιτικά ε, στοιχεία και τι μπορείτε να κάνετε, γιατί εσείς βλέπετε και τι ακριβώς συμβαίνει. Θα ήθελα λοιπόν ε, να ζητήσω από τους συναδέλφους ε, να κάνουν ερωτήσεις σε αυτή την κατεύθυνση και να μην ξεκινήσουν διάλογο. Να ξεκινήσουμε με τον εισηγητή, αν θέλετε. Τζιν, να ξεκινήσεις εσύ τη συζήτηση με τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σου και στη συνέχεια θα ακούσουμε τους υπολείπους. Τζιν. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ για την έκθεση και τα στοιχεία που μας δώσατε. Πολλοί από εμά νομίζω ότι θα συμφωνήσουν με αυτό που είπατε για την πτυχή της εφαρμογής. Δεν ξέρω αν μπορείτε να σχολιάσετε και λίγο περισσότερο τι γίνεται με το νέο τμήμα του κανονισμού του Δουβλίνου για την ε, ετοιμότητα και την ε, έγκαιρη προειδοποίηση του early warning. Αν ε, έχει γίνει δεκτό αυτό από τα κράτη-μέλη και να αρχίζουν να το εφαρμόζουν, διότι δόθηκε μάχη για να περάσουν αυτά. Όσον αφορά τώρα το ρόλο του Συμβουλευτικού Φόρουμ, μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια για το πώς χρησιμοποιείται αυτό πλέον και θα θέλαμε να μας απαντήσετε και το κατά πόσον Ενώ καλές, ε, αρκετές χώρες φαίνεται να έχουν αύξηση αριθμού αιτήσεων, φαίνεται να υπάρχει μία πτώση σε κάποιες χώρες, κατά την άποψή μου στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε αν υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό. Ευχαριστώ. Okay, thanks. Okay, the next one is... Ναι, ο κύριος Κίρκοπ. Τι αυτή. Θα είμαι πολύ σύντομο αυτή τη φορά κύριε Πρόεδρε, διότι τις γενικές πολιτικές παρατηρήσεις μου τις έκανα προηγουμένως. Τρία πράγματα να ρωτήσω προγράμματα περιφερειακής προστασίας. Είμαστε ικανοποιημένοι. Θεωρούμε ότι αυτά τα προγράμματα προστασίας με τρίτες χώρες έχουν κάποια αποτελέσματα. Εγώ δεν είμαι βέβαιος. Νομίζω ότι κάτι θα πρέπει να δούμε εδώ. Δεύτερον, όσον αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε μια κατάσταση ε, ενώπιον της οποίας επειδή δεν καταφέρνουμε να επεξεργαστούμε τα στοιχεία, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις αφήξεις στην πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, βλέπουμε αρκετούς ανθρώπους να μετακινούνται στην Ευρώπη σε αρκετές χώρες Έχουμε το πρόβλημα στο Καλέ ε, και από άλλες χώρες που δέχονται ε, μετανάστες τους οποίους δεν τους εξεργάζονται τις αιτήσει τους στη, χώρα πρώτης άφηξης. Μπορούμε να κάνουμε κάποια περισσότερα, να δοθούν κάποιοι περισσότεροι πόροι σε αυτές τις χώρες πρώτης άφηξης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ή επειδή δεν υπάρχουν κοινά πρότυπα σε χώρες ε, ε, ε και δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο οι άνθρωποι αυτοί, έχουμε τόσο μεγάλη μετακίνηση. Η κυρία Γκυγιόμ. Ευχαριστώ, θα είμαι και εγώ σύντομη για την έκθεση αυτή. Σα ευχαριστώ για την ποιότητα τη έκθεση. Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό το γεγονό και το είπατε κι εσείς ότι ε, θα πρέπει να έχουμε αυτή την οτροπία συνεργασία, η οποία θα πρέπει να αυξηθεί και να βελτιωθεί ε, στα κράτη-μέλη και μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την υπηρεσία σα. και φυσικά ε, αναφερθήκατε και στο ρόλο που έχει να διαδραματίσει η υπηρεσία. Μία παρατήρηση έχω να κάνω εδώ. Ε, η έκθεση είναι για την κατάσταση του ασύλου. Η έκθεση λοιπόν θα έπρεπε να μας επιτρέπει στο μέλλον να έχουμε μια πολύ καλύτερη ανάλυση ως προς τις προοπτικές του φαινομένου. Ε, υπάρχουν πολλές αναλύσεις και νομίζω ότι οι επικρίσεις θα έπρεπε να βοηθήσουν για να προχωρήσουμε και σε άλλα πεδία. Ένα αυτό και δεύτερον ε, θα ήθελα αν μπορείτε να μας πείτε δύο πράγματα για το τι ακριβώς ε, υπάρχει μεταξύ ε, της υπηρεσίας και κάποιων χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματος χάρη της Ελβετίας, αυτή έχω κατά νου, και να μας πείτε και δύο επιπλέον στοιχεία για τον προπολογισμό, γιατί αν κατάλαβα καλά η υπηρεσία ε, έχει διάφορες δραστηριότητες και φυσικά αυτό θα έχει συνέπειες και για το προσωπικό αλλά και για, το, για την ίδια την υπηρεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Φεράρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε συγκεκριμένα στα σχέσια στα πλαίσια του ειδικού προγράμματος στήριξης χωρών όπως η Ιταλία που δέχονται τις μεγαλύτερες ε, πιέσεις. Διότι αυτές είναι οι χώρες οι οποίες βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου αντιμετωπίζουν προβλήματα για να αντιμετωπίσουν ε, πολλές ε, διεθνεί αιτήσεις ασύλου και δεν μπορούν να σεβαστούν το χρόνο για να τηρήσουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ο στόχος ε, αυτής της προσφοράς ε, διεθνούς προσπασίας δεν είναι μόνο ε, για να γίνουν σε κατάλληλο χρόνο, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στην Ιταλία έρχονται άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν την ελευθερία τους και βρίσκονται υποκράτηση για μήνες μέχρι και ένα χρόνο, μέχρι να λάβουν καθεστώς πρόσφυγα. Και πολλές φορές βρίσκονται κρατούμενες σε μια χώρα στην οποία κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι ο στόχος τους. Ε, στα πλαίσια αυτών των μηνών, ε, ορισμένες φορές αναγκάζονται να ε, ζητιανεύουν και να κάνουν μικροεκκλήματα στους δρόμους. Απ' την άλλη υπάρχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι εξοργίζονται γιατί θεωρούν ότι γίνεται κακοδιαχείριση, ότι δεν γίνονται κατάλληλες επενδύσεις σε κοινωνικό επίπεδο, προκειμένου να βοηθήσουν τις χώρες να αντιμετωπίσουν καλύτερα την κατάσταση του ασύλου. Και πρόκειται για μια κατάσταση η οποία είναι αλυσιδωτή αντίδροση και επιμένω ως αυτό διότι δεν υπάρχει έγκαιρη ανταπόκριση, δεν υπάρχει σωστή απάντηση για διεθνή προστασία και δημιουργείται ένα αλυσιδωτό φαινόμενο το οποίο ε, στη συνέχεια οδηγεί σε ε, δυσπιστία ενώπιον των ξένων και ακόμα και διάκριση. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω και θα ήθελα να σας ρωτήσω πιο συγκεκριμένα τι ακριβώς είναι αυτό το ειδικό πρόγραμμα στήριξης για χώρες οι οποίες πιέζονται περισσότερο από τις μεταναστευτικές ροές. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Ντάλι, Μαρία. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τις πληροφορίες περί της υπηρεσίας. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το Λεάζο και εντυπωσιάστηκα. Ήταν πολύ θετική η εμπειρία. Λόγω όλων όσων έγιναν με τα περιορισμένα μέσα που διέθεταν. Ανησυχώ όμως για τους αριθμούς που υποβλήθηκαν σχετικά με τους αιτητές ασύλου. Το 13 ήταν έτος ρεκόρ και Νομίζω ότι το 2014 θα σημειωθεί νέο ρεκόρ. Μπορείτε να μας τα αποσαφηνίσετε κάπως καλύτερα. Διαπιστώνουμε πάντως ότι υπάρχει αύξηση του αριθμού ετητών ασύλου. Και αυτό πιέζει περισσότερο τα συστήματα υποδοχής, όπως λένε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκκλησή μου λοιπόν είναι να δώσουμε ένα σημαντικότερο ρόλο στο ΛΕΑΖΟ στην υπηρεσία της Μάλτας. Ο κύριος Γιούνκερ συνομίλησε με τον υποψήφιο επίτροπο για τα εσωτερικά και πρέπει να δούμε αν θα δοθεί περισσότερη σημασία σε αυτό το γραφείο υποστήριξης των, ε, των ασύλου και να δούμε αν θα έχει περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα να εφαρμοστούν πιλωτικά πειραματικά προγράμματα, ολόκληρα προγράμματα όμως, για τα σημαντικότερα θέματα, να αντιμετώπιση των σημαντικότερων θεμάτων, ας πούμε το joint processing. Και τώρα μερικά σύντομα ερωτηματάκια. Η δέσμη για το άσυλο που συζητήθηκε, θα ήθελα να ξέρω πώς, πώς, πώς πώς λέγω η δέσμη αυτή θα λειτουργήσει όπως πρέπει. Για το οργανωμένο έγκλημα και τη μετανάστευση θα ήθελα συγκεκριμένες πληροφορίες γιατί πολλές φορές μιλάμε για το φαινόμενο της, οργανωμένου εγκλήματος συνδεδεμένο με την μετανάστευση μόνο όταν σημειώνονται τραγωδίες όπως τη Λαμπετούζα και τη Μεσόγειο γενικότερα. Τέλος, το Γραφείο υποστήριξη στο ΛΕΑΖΟ για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του πρέπει να διαθέτει πόρους και την απαραίτητη εντολή. Να έχει το προσωπικό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του και τους πόρους το ξαναλέω και τους πόρους και τους πόρους Thank you. Uh, next is Scar Ευχαριστώ. Σκάκελερ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με το θέμα των πόρων. Το προσπαθούσαμε και πέρσι. Και βεβαίως και την εφαρμογή του πακέτου ασύλου. Υπάρχουν πολλά πράγματα, αν, δείτε, αν δει κανείς ε, την αναγνώριση ε, και την απόδοση ασύλου. Ε, πρώτα απ' όλα όμως ε, ο κ. Αβραμόπουλος ε, στην επιστολή του μας είπε πως θα πει, θα ζητήσει από την υπηρεσία σύλλου να συνεργαστεί με τρίτες χώρες, κάτι το οποίο για μας χτυπάει καμπανάκι. Γιατί βοηθάει υποτίθεται η διαδικασία σύλλου. Όχι να απομακρύνει τους ανθρώπους κάτι στο οποίο συνήθως στοχεύει συνεργασία με τρίτες χώρες. Μπορείτε να μας εξηγήσετε, έχετε κάποιες πληροφορίες για το τι σημαίνει αυτή η συνεργασία με τρίτες χώρες. Έχετε ιδέα για το τι πρέπει να κάνετε σε σχέση με τις τρίτες χώρες. Και ενδιαφέρον και αυτό το οποίο είπατε για το πιλωτικό έργο στη Μάλτα και την Ιταλία για τους λαθρεμπόρους. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει, ποιος είναι ο ρόλος σας και ειδικά αυτό με τις τρίτες χώρες. Μάλιστα. Όλοι είστε σύντομοι και σας ευχαριστώ. Λόπες Αγγιλάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Φίσερ για την παρουσίασή σας. Για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της υπηρεσίας σας, την οποία ξέρετε πως εκτιμώ. η Επιτροπή μας ε, ε ασχολείται με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ετούντων άσυλο η διεθνή προστασία στην πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. να κάνω μια ερώτηση που αφορά ένα θέμα το οποίο πάντα εμφανίζεται σε διάφορες διασκέψεις και αφορά τη λάθος αντίληψη που υπάρχει για την Ευρώπη. Τη λάθος αντίληψη. Είναι εντυπωσιακό να δει κανείς το πόσα λίγα ξέρει ο κόσμος για το γεγονότα για το άσυλο στην Ευρώπη. Ο κόσμος είναι πεπισμένος πως τα νότια κράτη-μέλη είναι γεμάτα ετούντες άσυλο. Αντιθέτως, οι περισσότερες αιτήσει είναι στη Γερμανία, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Σουηδία. Όχι ακριβώς οι πιο εκτεθειμένοι. Πώς ε, εξηγείται το φαινόμενο αυτό όσον αφορά την εφαρμογή ενός κοινού ε, συστήματος ε, ασύλου. Γιατί δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την νομική σφαίρα. Υπάρχουν ε, διεθνείς συμβάσεις της Γενέβης, το πρωτόκολλο 51-67 της Νέας Υόρκης. Better, how can we better report and inform πώς θα ενημερώσουμε και θα διαδώσουμε τα πραγματικά γεγονότα. Και η δεύτερη μου ερώτηση, πώς θα εξηγήσουμε και πώς εξηγούμε αυτές τις τεράστιες διαφορές στην εφαρμογή κανόνων που υποτίθεται πως είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα. και δεύτερον πώς θα φροντίσουμε ο κάθε ένας που κάνει αίτηση για άσυλο να έχει τουλάχιστον την ευκαιρία να έχει τουλάχιστον μια ευκαιρία Αναφέραμε εδώ στην αρχή της ε, μη επαναπροώθησης, ε, ε π.χ. όταν ε, λαμβάνουμε κάποιους ε, προφανώς παράτυπους μετανάστες στην, στην ξηρά, δηλαδή στη Θεούτα, τη Μελίγια, στις παραλίες της Ισπανίας ή και στη Μάλτα ή στα νησιά της Ελλάδας ή στη Λαμπεντούζα ή τα άλλα νησιά της Ιταλίας. Όταν υπάρχει εκεί πέρα κάποιος ο οποίος θέλει να ζητήσει άσυλο, να έχει τουλάχιστον μια ευκαιρία. Γιατί έτσι που κάνουν τα κράτη-μέλη, ε, τους βάζουν σε κάποιο κέντρο, όπως και αν το λένε, και εφαρμόζουν συνθήκες επαναπατρισμού με χώρες ε, συνορικές, ε, με χώρες ε, γειτονικές ή με χώρες προέλευσης ή αυτές που υποψιαζόμαστε ότι είναι. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. όταν ε, έχουμε ακριβώς και κάποια σημεία ιδιαίτερης έντασης του φαινομένου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εγώ κατάλαβα τι λες. Πράγματι. Βλέπουμε πως ε, τα νούμερα για Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο είναι σχετικά υψηλά, αλλά προφανώς ε, η αντίληψη που υπάρχει είναι γιατί πρώτα στις νότιες χώρες πάνε, ε, βλέπει κανείς που είναι η πίεση αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λες. Και σε ευχαριστώ. Κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για την έκθεση, κύριε Βίσερ. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Επειδή η επιχείρηση Mare δεν θα αντικατασταθεί από τη Frontex ε, ΣΥΝ, και υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες για τη φορονταξίν, για την χρηματοδότηση και για τις ε, πραγματικές διαστάσεις επιχείρησης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορούμε να προβλέψουμε ίσως και την παρουσία ενός ε, υπαλλήλου της ΕΑΣΟΥ σε σε οποιαδήποτε ε, επιχείρηση αναζήτησης και διάσωσης της Frontex, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι προστατεύονται πάντα τα δικαιώματα των ετούντων άσολο. Σας το λέω αυτό διότι υπάρχει μια συμφωνία του 2012 μεταξύ ΕΑΣΟ και Frontex και επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι δυστυχώς υπάρχουν χώρες, μεταξύ των οποίων και η δική μου, η Ιταλία, στην οποία δικαίως ε, γίνεται συζήτηση και εγώ γίνω μάχη ε, γι' αυτό για να καταπολεμήσουμε την παρανομία και το οργανωμένο έγκλημα αλλά στην ε, διαδικασία αναζήτησης και διάσωσης που κάνουν τα σκάφη πολύ συχνά διασώζονται άνθρωποι από ναυάγια οι οποίοι τιμωρούνται στη συνέχεια και ε, διώκονται ποινικά, νομικά επειδή διέσωσαν ανθρώπους στη θάλασσα. Ευχαριστώ. Η κυρία Στίβενς. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον βλέπω πως ε, έχουν δικαίωμα όσοι ζητάνε άσυλο στη διερμηνία. Υπάρχει στην Αλλά ε, έχω κάποιες ερωτήσεις ε, ε, όσον αφορά τη διερμηνία σε άτομα τα οποία δεν ακούνε. Πώς θα διασφαλίσουμε πως ε, οι κοφοί οι οποίοι κάνουν αίτηση ασύλου θα έχουν ποιοτική διερμηνία. Ε, βεβαίως θα είναι προφανώς με τα, με τα σύμβολα. Το θέμα είναι σε ποια γλώσσα θα είναι η ε, διερμηνία προς ε, κουφούς και βεβαίως και το ζήτημα ευπαθών ατόμων, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θετικό. Γιατί υπάρχει εδώ πέρα κίνδυνος κατάχρησης. Βλέπουμε στο Βέλγιο άτομα με αναπηρία τα οποία εξαναγκάζονται να ζητιανεύουν που είναι ένα άλλο πρόβλημα μετά αλλά θέλω να θέσω το ερώτημα Έχετε σκεφτεί καθόλου να αφιερώσετε κάποιους πόρους για λεσβίες και τρανσέξουαλ καθώς επίσης ε, και γυναίκες οι οποίες εξαναγκάζονται σε πορνεία ή έχουν ακροτηριαστεί. Γιατί δεν βλέπω εδώ πέρα τίποτα για ιδιαίτερες ομάδες για ε, ανάπηρους ειδικά. Σκοπεύει λοιπόν η Κομισιόν να κάνετε κάτι τους επόμενους μήνες ε, ειδικά για τα άτομα με αναπηρία ε, γιατί και εκεί πέρα όταν μιλάμε αναπηρίες υπάρχουν πολλές κοφοί, τυφλή οι άνθρωποι με νοητική υστέρηση είναι πολύ ευπαθείς ομάδες τους λαμβάνετε υπόψη. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Thank you very much, Stevens. I think we were just... Ευχαριστούμε πολύ κυρία Stevens. Έχουμε ακόμη μακρύ κατάλογο. Αν θέλει κανείς άλλος να μιλήσει να το δηλώσει τώρα. Εσείς είστε στο κατάλογο. Άλλος, άλλος, άλλοι. Δύο ακόμα. Μάλιστα. Ξέρετε τι λένε στους γάμους. Τώρα να τα δηλώσετε αλλιώς. προειδοποίησα τον Ροβέρτο ότι θα υπήρχαν πολλές ερωτήσεις. Ο κ. Σταντόσκι τώρα. Σε τι γλώσσα θα μας μιλήσει σήμερα. τσεχικά σήμερα. ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ και για την ε, εξαιρετική έκθεση. Πολύ ωραία με τα διαγραμματά της, ε, κύριε Φίσερ, ε, μία από τις ωραιότερες εκθέσεις που έχουμε δει. τον καιρό τουλάχιστον που είμαι εγώ ευρωβουλευτής. Σας βγάζω το καπέλο λοιπόν. Κοιτάξτε, εμένα με ενδιαφέρουν οι Ρώσοι που ζητάνε άσυλο στην Τσεχία. Έχουμε πολλούς Ρώσους, ε, πολλοί έρχονται σε μας, κυρίως λόγω της ε, καταπίεσης ε, του καθεστώτος Πούτιν ε, σε όσους δεν είναι υπέρ του καθεστώτος. Παραδείγματο χάρη δημοσιεύτηκε κατάλογος των ατόμων που πέθαναν οι γη τους στην Ουκρανία και άλλα τέτοια. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις ε, ανθρώπων από την Τσετσενία. Άνθρωποι που τιμωρήθηκαν για πράξεις ε, που δεν είναι αξιόπινες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή το πολύ πολύ να πλήρωναν πρόστιμο, ξέρω εγώ. Ξέρουμε πώς είναι αυτές οι περιπτώσεις. Στον τομέα αυτών λοιπόν σχεδιάζεται να υπάρχει κάποια μεγαλύτερη ευελιξία γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Σας ευχαριστώ κυρία Βερζία. Ε, μιλήστε όσο θέλετε. Δώστε του να καταλάβει. Όχι, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου. Συμφωνώ με όσα υπόθηκαν για την ποιότητα της έκθεσης γιατί πράγματι είναι πολύτιμο εργαλείο ανάλυσης. Θέλω όμως να τονίσω το εξής, να προσέξουμε και εμείς και άλλοι τη χρήση αυτών των ξερών στατιστικών στοιχείων. 77% λέει, μιλάει για 100 και για άλλα ποσοστά, τι παιχνίδι είναι αυτό, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι αριθμοί από ορισμένους, το βλέπουμε ήδη από δημοσιογράφους, είναι επικίνδυνο και δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα εκείνων που θέλουμε να προστατεύσουμε. Αυξήσεις 700% είναι κάτι που πρέπει να σχετικοποιηθεί σε σχέση με τα πραγματικά ποσά και οι αριθμοί αυτοί έτσι χωρίς ανάλυση είναι ανησυχητική. Επίσης πρέπει να τονίσουμε τις διαφορετικές καταστάσεις που ισχύουν για πολλούς αιτητές ασύλου και τον τρόπο με τον οποίο τους μεταχειρίζονται τα κράτη-μέλη. Και πριν και μετά την αποδοχή του αιτήματός τους εμένα με εντυπωσιάζει η αύξηση του ποσοστού ενδιάμεσης θα έλεγα προστασίας έναντι του πραγματικής κατάστασης του καθεστώτος του ασύλου. Μήπως τελικά μειωθεί η προστασία από το ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση των καθεστώτων ή της νομοθεσίας. Επίσης αναρωτιέμαι και κάτι που δεν τονίζεται αρκετά στην έκθεση το θέμα της χώρας προορισμού και του πραγματικού προορισμού αυτού που ζητάει το άσυλο ας πούμε το καλέ 2.000 αλλά γιατί υπάρχει αυτός ο θύλαξ εκεί στο Καλέ διότι έρχονται αγγλόφωνοι από χώρες της Ανατολικής Αφρικής μιλάνε αγγλικά δεν θέλουν λοιπόν να παραμείνουν τελικά ούτε στην Ιταλία ούτε στη Γαλλία ούτε στην Ελλάδα αν αυτό δεν το δούμε δεν θα καταλάβουμε Χρειάζεται λοιπόν μία αντιμετώπιση πιο σφαιρική. Και ξαναλέω για την Ερυθρέα γιατί δεν ήταν ικανοποιητική η απάντηση. Πρέπει να το ξαναδούμε και να προσέξουμε επίσης επειδή συνάντησα χθες Ερυθρέους τα λέω αυτά δύο παραδείγματα τι μας είπαν σε κάποιο γραφείο ασύλου ζήτησαν από έναν να υποβάλει τα διπλώματά του στο, από την πρεσβεία αλλά με αποδεικτικά στοιχεία πλήρη και ο άλλος μας μίλησε για τις συνθήκες κράτησης ή διαβίωσης στην Ερυθρέα γιατί η Ερυθρέα είναι ολόκληρη σαν υπαίθρια φυλακή. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια προσπάθεια εδώ. Ευχαριστώ. Δεν θα ήθελα να χάσω άλλους συναδέλφους γιατί είναι σημαντικό θέμα και θα ήθελα να έχουμε αρκετές ε, σημαντικές απαντήσεις από τον κύριο Βίσερ. Θα ήθελα από τους επόμενους να ζητήσω να περιοριστούν στο ένα λεπτό ε, ιδίως αν ε, μίλησαν στην προηγούμενη συζήτηση. Σας παρακαλώ να είστε όσο το δυνατόν πιο σύντομοι. Ο κύριος Μπέκερ από το ΕΛΚ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Ανάφερε ο κύριος Φίσερ πως η έκθεση εδώ πέρα οπωσδήποτε ε, καταρτίστηκε γνωρίζοντας τα γεγονότα του 2013. Αναφέρομαι εδώ πέρα στο θέμα του κώδικα ε, της ε, βίζας. Ποιες συγκεκριμένες προγνώσεις έχετε όσον αφορά την ανανέωση του κώδικα θεωρήσεων αφενός και αφετέρου για την ε, βίζα αυτή επιστροφής γιατί θα ήθελα να πω πως ο αριθμός αυτών των θεωρήσεων είναι κάτι το οποίο εγώ βλέπω κάπως επιφλεκτικά αλλά ε, χαιρετίζω την πρωτοβουλία σας αλλά θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η πρόγνωσή σας τι μπορούμε να περιμένουμε ως Ευρώπη ευχαριστώ ευχαριστώ Κοράω Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα είμαι πολύ σύντομος ήθελα απλώς ε, να ρωτήσω από τον κύριο Βίσερ από την υπηρεσία Εάν είστε ικανοποιημένοι από την εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου, εάν θεωρείτε ότι ο κανονισμός του Δουβλίνου απλώς επισημαίνει το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένωση στην ένωση. Διότι είναι σαφές ότι εάν σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου εμείς πάντα χρησιμοποιούμε τη διακυβερνητική μέθοδο και όχι την κοινοτική μέθοδο, οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, θεωρούν ότι η Ένωση αυτή όταν ε, αφορά τέτοια θέματα δεν υπάρχει. Και το θέμα απλώς επαφίεται στα κράτη-μέλη τα οποία ε, υποδέχονται μεταναστευτικές ροές πολύ πιο μεγάλες σε σχέση με άλλες χώρες. Και επίση, όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα στήριξη στην Ιταλία, το οποίο ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του 2014, υπάρχει πρόθεση παράτεσή του. Ευχαριστώ. Thank you. And Mrs. Ευχαριστώ, κυρία Κανίτσι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Βίσερ για την έκθεσή σας, η οποία είναι πληρέστατη και μας παρουσιάζει τα όσα έκανε η Άσο. Η κατάσταση όμως που μας παρουσιάζεται στην έκθεση δεν θα πρέπει να το κρύβουμε άλλωστε, είναι ανησυχητική. Έχουμε αύξηση των μεταναστευτικών ορών ε, κατά 30% και των αιτήσεων ε, ε, προστασίας. Μήπως θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν λοιπόν από την έκθεση συμπεριλαμβανομένων και αυτά για το ποσοστό αναγνώρισης ε, ε, σε σχέση με τις ε, ροές και τον, τα κράτη τα οποία ε, επεξεργάστηκαν τις αιτήσει ασύλου σε τρεις πτυχές. Καταρχάς να υπάρχει μεγαλύτερη δέσμευση για να μπορέσουμε να προλάβουμε και να διαχειριστούμε αυτές τις ροές οι οποίες όπως αποδεικνύεται από την έκθεση σχετίζονται με κρίσιμες καταστάσεις όχι σε όλο τον κόσμο αν μου επιτρέπεται η, έκ, έκφραση αλλά κυρίως στα σύνορα ή κοντά στα σύνορα της Ένωσης. Τα Βαλκάνια, η Συρία, ο Κάφκασος και όπως υπογραμμίζει είστε και εσείς προηγουμένως, προσφάτως και Ουκρανία. Ε, επίσης, αν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία, θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την εναρμόνιση στα κράτη-μέλη του συστήματος του Δουβλίνου ε, και σε σχέση με τα ε, αιτήματα μετεγκατάστασης. Και αυτό για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ομογενή κατανομή και επομένω και πιο διαχειρίσιμη στα πλαίσια καλύτερης ένταξης ε, για τους αιτήντες άσυλο και ξέρουμε ότι κυρίω τους υποδέχονται κυρίω στη Γερμανία, στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σουηδία και στη χώρα μου, στην Ιταλία. Και τέλο, θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία για μείωση του χρόνου εξέταση των αιτήσεων που ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη κυρίω όσον αφορά κάποιε χώρε και κάποιε συγκεκριμένε ε, ε, ροέ. Και τέλο, ε, κατά πόσο θα μπορούσαμε να τελειοποιήσουμε και το μηχανισμό έγκαιρη προειδοποίηση και προετοιμασίας και διαχείρισης της κρίσης που προβλέπεται από το άρθρο 33 του νέου κανονισμού του Δουβλίνου. Και τέλος, και με αυτό ολοκληρώνω, αν μπορείτε να μας δώσετε κάποια επιπλέον πληροφορία για τα όσα ξεκινήσατε με τη Eurojust και τη Europol για να αντιμετωπίσετε τις κλιματικές οργανώσεις οι οποίες ε, ε, διαχειρίζονται την ε, εμπορία ανθρώπων. Ευχαριστώ. Η κυρία Μέτσολα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε δύο ερωτήσεις και θα είμαι και σύντομη. Όσον αφορά την ε, μετεγκατάσταση, θα ήθελα να συνεχίσω με αυτό που είπα προηγουμένως. Η μετεγκατάσταση μειώθηκε. Και ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι το Νοέμβριο θα γίνει ένα ετήσιο φόρουμ για τη μετεγκατάσταση. Το έχουμε συζητήσει αυτό, κύριε Βίσερ, αλλά θα ήθελα να επισημάνω το εξή. Στην ε, εντολή της ΕΑΣΟ υπάρχει συγκεκριμένος ρόλος για τα θέματα μετεγκατάστασης και εγώ περιμένω από την ΕΑΣΟ να έχει πιο δραστηριό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα τις ανησυχίες και τις δυσκολίες ε, των κρατών μελών, ώστε να μπορούν να αποδεχτούν αυτή την έννοια, ότι πρόκειται για κάτι το οποίο είναι θελοντικό, το οποίο έχει αποτελέσματα και το οποίο είναι ένδειξη αλληλεγγύης. Δεύτερον, όσον αφορά την Task Force για τη Μεσόγειο και το πρόγραμμα δράσης της ΕΑΣΟ. Στην έκθεση αναφερθήκατε σε αυτό και είπατε, λέει μάλλον η έκθεση, ότι όλα αυτά γίνονται υπό όρους και ότι μπορεί να έχει περισσότερη σχέση με συγκεκριμένε χώρες. Μπορεί να υπάρχουν προγράμματα προστασίας, για παράδειγμα, στη Λιβύη. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω γι' αυτό. Ποιοι είναι οι στόχοι της ΕΑΣΟ, ώστε να μην ε, βλέπουμε απλώς το κείμενο για την ετήσια έκθεση, αλλά να υπάρχει και κάποια παρακολούθηση για τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κέγκε. Sí. Ναι, ευχαριστώ ευχαριστώ και από πλευράς μου για την έκθεση η οποία μας επιτρέπει να αντιληφθούμε λίγο καλύτερα και το θέμα και το τι ακριβώς κάνετε. Η ερώτησή μου θα είναι αρκετά σύντομη. Από ό,τι είδα υπάρχει οδηγία του 2001, η οδηγία 55 του 2001, η οποία αναφέρεται στους ελάχιστους κανόνες για το προσωρινό καθεστώς προστασίας σε περίπτωση που υπάρχει μαζική εισρωή και φυγή από κάποιες χώρες. Μέχρι τώρα όμως επαφίεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει ε, έναν αριθμό για το κατά πόσο θα πρέπει να εφαρμόζεται αυτό. Μήπως θα έπρεπε να επανεξετάσουμε τα αριθμητικά κριτήρια για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας, η οποία περιλαμβάνει πολλά στοιχεία, τα οποία κατά την άποψή μου θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στα κράτη-μέλη, ώστε να ε, έχουμε πραγματικά αλληλεγγύη και συνεργασία, που βλέπω ότι περιλαμβάνονται ως κριτήρια σε αυτή την οδηγία. Η δεύτερη ερώτησή μου είναι η εξή. Βάσει της ανάλυσης που μας κάνατε, μήπω θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να επαναξετάσετε τα κριτήρια για το ε, για τον καθορισμό του νομικού καθεστώτος, διότι εξετάζοντας απλώς τη χώρα καταγωγής ε, κάποιου ο οποίος κάνει αίτηση ασύλου, ε, μπορεί κάποιος να μην προέρχεται από μια χώρα στην οποία υπάρχει ένοπλη σύραξη, αλλά να προέρχεται από κάποια χώρα στην οποία να υπάρχει πολύ μεγάλη ξηρασία. Μήπως θα έπρεπε να επανεξετάσουμε λοιπόν και τον καθορισμό των διαφόρων κατηγοριών προσφύγων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τέλος, η κυρία Σλάιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Βίσερ για την έκθεση. Ε, το είπαν αρκετοί. Οι μεγάλες αστάθειες ε, γύρω από τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή ε, συνεισέφεραν σημαντικά στις μεταναστευτικές ροές της Ευρώπης και κυρίως στις χώρες ε, που βρίσκονται ε, στα σύνορα, στα, στα νότια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν μεγάλε μεταναστευτικέ ροέ και είναι πολύ σημαντικά τα προβλήματα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα όλων και από εκεί και πέρα ε, θα πρέπει να καθορίσουμε και το νομικό μα καθήκον. Δεν φτάνει το ηθικό μα καθήκον να σώσουμε οποιονδήποτε ξεφεύγει από πολέμου, από βασανισμού ε, ή από πολύ επικίνδυνε καταστάσει. Επειδή η Μεσόγειο, που είναι μια ευρωπαϊκή θάλασσα, γίνεται χώρο ε, τραγωδία και θανάτου, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βίζερ μήπω θεωρεί ότι θα ήταν καλύτερα να έχουμε κάποιε λύσει οι οποίε να προλαμβάνουν τι παρεμβάσει. Παραδείγματο χάρη ασφαλεί λιμένε, του οποίου θα μπορούσε κάποιο να ζητήσει προστασία στι χώρε τη διέλευση με ε, διεθνή προστασία, ώστε ακριβώ να μην φτάνουν ε, οι ε, μετανάστε στα χέρια των εμπόρων που του αφήνουν να πεθάνουν στη θάλασσα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βίσερ, να σας δώσουμε το λόγο Έχουμε μία σειρά από διάφορες ερωτήσεις, πολιτικές, επιχειρησιακές, νομικές και σας παρακαλώ να απαντήσετε όσο καλύτερα μπορείτε γιατί είναι και, μεταδίδεται και ζωντανά στο διαδίκτυο η Επιτροπή. Έχετε όσο χρόνο θέλετε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους βουλευτές. Εντυπωσιακό ο κατάλογος εδώ πέρα. Για ένα θέμα πολύ σημαντικό. Οπότε χαίρομαι και για τις ερωτήσεις και για τη δυνατότητα που έχω να απαντήσω. Υπάρχουν κάποια πράγματα ε, τα οποία συμφωνείτε και κάποιες πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω πολύ συγκεκριμένα. Αν μου ξεφύγει κάτι θα είναι κατά λάθος, σας διαβεβαιώ. Να ξεκινήσω με την ετήσια έκθεση και το τι εννοούμε. Να μπορούμε να ερμηνεύσουμε το μέλλον, αν υπάρχουν κάποιες προειδοποιήσεις, πώς θα είμαστε έτοιμοι όλα αυτά νομίζω συνεισφέρουν. Εγώ πιστεύω πως ε, μια ευρωπαϊκή υπηρεσία πρέπει να έχει κάποια προσθέμενη αξία, Αλλιώ να την κλείσουμε. Αυτό το οποίο βλέπουμε λοιπόν είναι ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται σε τομείς ε, όπου μέχρι τώρα δεν είχαμε την ε, δυνατότητα. Αυτό ξεκινάει με ε, δεδομένα και πληροφορίες. Ο κύριος Λόπελ Ζαγγιλάρ ε, τοποθετήθηκε επί της αρχής στο όλο ζήτημα έκανε μία σύνοψη και είπε ουσιαστικά σωστά ερμηνεύουμε τα πράγματα αν πως υπάρχουν κάποιες λανθασμένες αντιλήψεις και αν μπορούμε να έχουμε καλύτερα ε, στοιχεία για να γίνει μια κάπως διαφορετική συζήτηση. Ως ένας ταπεινός εκτελεστικός διευθυντής, ε, εγώ θεωρώ πως καθήκον μου είναι ε, να σας δώσω τα στοιχεία. Και, ναι, υπάρχουν πολλές λάθος ιδέες. Δεν θα αρχίσω εγώ τώρα να τις αναφέρω γιατί θα ξεκινήσει μια συζήτηση που δεν θα τελειώσει ποτέ αλλά είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Αυτή είναι νομίζω η βασική συνεισφορά μιας ετήσια έκθεση. δηλαδή από χρόνο σε χρόνο να σας δίνουμε τα δεδομένα για να τα χρησιμοποιήσετε εσείς ως πολιτικοί και να πείτε ίσως πρέπει να αλλάξει αυτό Ίσως εάν αυτά είναι τα πραγματικά στοιχεία, αν αυτή είναι η πραγματικότητα, τότε μπορούμε να αλλάξουμε το μήνυμά μας, να αλλάξουμε την ομοθεσία. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι στα χέρια σας. Πολύ πρακτικό επίσης. Ποιο είναι το κομμάτι που αφορά την έγκαιρη προειδοποίηση. Ξεκινήσαμε πριν από δύο χρόνια να ζητάμε από τα κράτη-μέλη να μας δίνουν δεδομένα σε αιτήσια βάση έτσι ώστε από μήνα σε μήνα να βλέπουμε τις αλλαγές, τις τάσεις στα κράτη-μέλη και στο σύνολο. Το δημοσίευμα ανατρίμηνο η, η μηνιαία έκθεση δεν δημοσιεύεται δυστυχώς, ίσως κάποτε να δημοσιεύεται και αυτή γιατί είναι σημαντικό να δούμε ποια είναι η τάση που υπάρχει. Και εδώ συμφωνώ και διαφωνώ με την παρατήρηση για τα ποσοστά. Συμφωνώ πως τα ποσοστά μπορούν να ξεγελάσουν και να αποπροσανατολίσουν. Ταυτόχρονα σε καθημερινή επιχειρησιακή βάση χρειάζεται μια απάντηση στο ερώτημα αν υπάρχει αλλαγή, αν προς τα που κινούνται οι τάσεις για πρακτικούς λόγους, για πρακτικούς λόγους με συγχωρείτε, ε, τα κράτη-μέλη πρέπει να οργανωθούν. <laughs> Οπότε αν έχουμε μια αύξηση 600% ε, και από χαμηλή εκκίνηση, ε, κάτι σημαίνει αυτό που αφορά και το Υπουργείο Οικονομικών. Έτσι. Πρακτικά πράγματα, αλλά με συγχωρείτε έτσι είναι η πραγματικότητα. Οπότε θα είμαστε πολύ προσεκτικοί με τα ποσοστά δεκτών, αλλά δεν είναι δυνατόν να εργαστούμε χωρίς νούμερα. Έγκαιρη προειδοποίηση. Από όταν ξεκινήσαμε, έχει γίνει ένα μέσο για τα κράτη-μέλη, την Κομισιόν και για εμάς ε, για να είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κανένα μεμονωμένο κράτος μέλος δεν είχε διαπιστώσει κάποια εισρωή από την Ουκρανία, αλλά εμείς το παρατηρήσαμε και είπαμε πως πρώτον δεν είναι τα κράτη-μέλη μόνο τους, δεύτερον να προετοιμαστούν γιατί δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, αλλά είναι κάτι το οποίο ε, είναι μια σοβαρή κατάσταση. Το ίδιο με το Ιράκ και τη Συρία. Ένα πρακτικό μέσο λοιπόν με προσθέμενη αξία. Επίσης υπάρχει ένα ενδιαφέρον νέο φαινόμενο που δεν είχαμε συνειδητοποιήσει. Αν δούμε τους Ερυθρέους. Συνολικά είδα μια μεγάλη αύξηση και ακόμα αυξάνε το αριθμός. Αλλά βλέπουμε πως οι ε, ομάδες τους, ε, γιατί είναι ομάδες, αλλάζουν από χώρα σε χώρα. Κράτη-μέλη που είχαν ε, αύξηση 800% και μετά από δύο μήνες ξανάψαν σε πολύ χαμηλά νούμερα και ξαφνικά βλέπουμε τα νούμερα να ανεβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος. Και συνειδητοποιούμε, βεβαίως όταν συνειδητοποιούμε ότι το σύνολο εξακολουθεί να αυξάνεται, ξαφνικά είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει. Η Ερυθρέα. Ελπίζω να μην παρεξηγήσατε δεν ξε... Όταν είπα δεν ξέρουμε τους λόγους, ε, εντάξει, ο ε, αριθμός ε, απόδοσης σύλλου είναι πάρα πολύ υψηλός. Οπωσδήποτε δεν υποτιμάμε την κατάσταση στη χώρα, αλλά τούτου λεφέντος καλό είναι να δούμε το φαινόμενο σε βάθος να δούμε και τους λόγους για να αντιδράσουμε καλύτερα. το Συμβουλευτικό Φόρουμ. Είναι ο οργανωμένος διάλογος με την κοινωνία των πολιτών. Πέρσι, μόνο πέρσι είχαμε 70 επαφές παρεμβάσεις με ΜΚΟ μέρος της εργασίας μας. Ζητούσαμε τη συμβουλή τους και βεβαίω ε, παραμένουν αυτοί υπεύθυνοι από τη δικιά τους την πλευρά εμείς από τη δικιά μας αλλά ε, υπάρχει μια αλληλεπίδραση με την κοινωνία των πολιτών και μάλιστα μετά από την συνεδρίαση εδώ πέρα θα συνεδριθώ με την ε, συμβουλευτική ομάδα του Συμβουλευτικού Φόρουμ Οπότε κάθε μέρα με αυτό το θέμα ασχολούμαστε. Τώρα, να δω κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Άτε. Περιφερειακά προγράμματα προστασίας. Να το πω ευρύτερα, γιατί υπάρχουν διάφορα ερωτήματα για τις εξωτερικές σχέσεις λοιπά ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος μας εδώ πέρα. Κοιτάξτε. Εγώ επιφυλακτικά το βλέπω γιατί ε, υπάρχουν ε, πολλοί τομείς ε, πολιτικής που αφορούν τον υπόλοιπο κόσμο. Αναπτυξιακή βοήθεια, εξωτερική πολιτική κτλ. Η μετανάστευση είναι μόνο ένας τομέας. Βεβαίως, εμείς τον θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό, αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. ρεαλιστές. Και... Κοιτάξτε, είναι χρήσιμο να κινητοποιηθούμε μόνο όταν μπορούμε να έχουμε προσθέμενη αξία, αλλά ε, δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο από τη σκοπιά της μετανάστευσης. Οπότε πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ε, και έτσι ερμηνεύω και τις παρατηρήσεις του νέου πρόεδρου της Κομισιόν για τον ρόλο της υπηρεσίας μας και την εξωτερική διάσταση. Δεν θα πάμε να αλλάξουμε την Αφρική ούτε να γίνουμε γραφείο στήριξης της Αφρικής. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Αλλά οπωσδήποτε σε πολύ συγκεκριμένα έργα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τις δυνατότητες της διοίκησης σε συγκεκριμένε χώρες. Τώρα δεν ξέρω αν η Λιβύη αυτή τη στιγμή είναι η πιο εύκολη περίπτωση. Αλλά εάν δείτε την Τινησία, την Ιορδανία, το Μαρόκο, οπωσδήποτε εκεί μπορούμε να εργαστούμε με τρόπο θετικό για να ενισχύσουμε την αποστολή μας. Ε, επίσης όσοι ζητάνε άσυλο και πάνω από τη μια χώρα στην άλλη. Πολλοί το, ναι, το περιγράφουν αυτό ως shopping ασύλου, αλλά είναι απλώς ένας τρόπος να δει κανείς το πρόβλημα στο κανονισμό του Δουβλίνου πολλά χρόνια ήδη πριν προσπαθήσαμε να μειώσουμε τον αριθμό αυτό ανθρώπων που κάνουν shopping ασύλου, ψώνισμα ασύλου οι λόγοι για τους οποίους μετανάστες πηγαίνουν σε κάποια χώρα είναι πολλοί. Μπορεί να είναι η γλώσσα, η ιστορία, η οικογενειακή λόγοι, σχέσεις με κοινότητες, ας πούμε για την Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει πολλούς, στέλνει πολλούς μετανάστες σχεδόν σε όλες τις χώρες της νόμιμους μετανάστες που έχουν δουλειά και που απλώς μετινάστευσαν όπως και πολλοί από εμά στο παρελθόν. Αλλά όταν γίνονται γεγονότα σαν αυτά τα τελευταία της Ουκρανίας μπορεί να υπάρχει και λόγος ότι έχουν γνωστούς και προτίθενται και άλλοι μετανάστες. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι μετανάστες πηγαίνουν σε κάποια χώρα. Τους αναλύουμε όλο και περισσότερο και ελπίζουμε σε σύντομα να μπορούμε να σας δώσουμε περισσότερες αναλύσεις για αυτό το σημαντικό θέμα με βάση αριθμούς και στοιχεία. Και φυσικά υπάρχουν και πολιτικά θέματα. Πολιτικά αλλά σας υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχετε την πληροφόρηση που χρειάζεστε. Για Αυτό απαντά και το θέμα των σχέσεων με γειτονικέ χώρες. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. αν οι μετανάστες πάνε κατευθείαν από ένα μέρος εκτός Ένωσης προς την Ένωση πρέπει να περάσουν σύνορα. Και οι χώρες είναι όλες χώρες σύνορων αφού έχουν αεροδρόμια αλλά μερικές έχουν και λιμάνια και βρίσκονται και στα εξωτερικά χερσαία σύνορα. τον μεγάλο αριθμό αιτητών ασύλου που έρχονται νομίμως, με νόμιμα μέσα που έχουν θεώρηση που ήταν φοιτητέ, ας πούμε ένας Ιρακινός φοιτητή από εκεί που δρά το Χαλιφάτο. Είναι κατανοητό να ζητήσει αυτός άσυλο. Δεν είναι αλήθεια λοιπόν ότι όλοι οι αιτητές ο συνολικός αριθμός που βλέπετε στην έκθεση για φέτος, ότι όλοι δηλαδή τους τελευταίους μήνες, εβδομάδες, ήρθαν μέσω διέλευση συνόρων. Μπορεί να έχουν έρθει με διαφορετικό τρόπο και με διέλευση συνόρων βέβαια και, αλλά να μην το ξεχνάμε. ειδικό υποστηρικτικό πρόγραμμα για την Ιταλία στοχεύει έχει στόχους προσαρμοσμένους στα προβλήματα της χώρας αυτής ως προς τη διαδικασία χορήγησης ασύλου για τις πληροφορίες που ζητιούνται για τη χώρα προέλευσης, την εφαρμογή του συστήματος του Δουβλίνου, για τα στατιστικά στοιχεία, Η Ιταλία είναι ομοσπονδιακή χώρα και έχει διαφορετικές παραδόσεις από άλλες ως προς τη διεκπαιρέωση τέτοιων και συλλογή τέτοιων πληροφοριών. Το πρόγραμμα τελειώνει φέτος και αυτή τη στιγμή το συζητάμε το μελλοντικό ένας συναδελφός μου είναι στη Ρώμη τώρα για την επέκταση, η παράταση του ή για ένα νέο τελείως πρόγραμμα από του χρόνου. Και επειδή η κατάσταση στη Μεσόγειο είναι αυτή που είναι, θελήσαμε να δούμε και πώς θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την Ιταλία λόγω το χρονο και επειδη αριθμού προσφύγων που έρχονται από τη Μεσόγειο. εφαρμογή της δέσμης ασύλου. Όλοι λένε ότι πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στη σωστότερη εφαρμογή αντί σε νέα μέτρα. Αυτό λέμε κι εμείς για το χρόνο και τώρα χωρίς να ξεχάσουμε βέβαια το γεγονός ότι η μετανάστευση είναι δυναμικό φαινόμενο και ότι οι σημερινές λύσεις δεν πρέπει να είναι πάντα και οι αυριανές. Προσέχουμε λοιπόν και αυτό το θέμα. Η εφαρμογή λοιπόν εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική γιατί πρέπει να εκπαιδευτεί το προσωπικό για τη νέα δέσμη ασύλου, για τη νέα νομοθεσία. Για να φανεί ότι είναι πιο αποτελεσματικό το ενιαίο e σύστημα από 27 διαφορετικά. Επίσης τέθηκαν ερωτήματα για σχέδια με τη Μάλτα και την Ιταλία για το φαινόμενο του λαθρεμπορίου. ή όπως λέμε εμείς για τη διευκόλυνση των οργών στη Μεσόγειο. In its actual that το πρόγραμμα αφορά ακριβώς αυτό το φαινόμενο, όχι με μονομένες περιπτώσεις ατομικές. Γιατί θέλουμε να συλλεχθούν πληροφορίες που μέχρι τώρα δεν είχαν συλλεχθεί. Έτσι ώστε όποιος έχει έρθει με κάποιο πλοίο να σκεφτούμε αν έχει επαφές με κάποια ενιαία οργάνωση δεν μπορεί να είναι όλοι από διαφορετική προέλευση ποιοι λοιπόν διευκολύνουν το λαθρεμπόριο μεταναστών αυτά βέβαια με στοιχεία ανώνυμα και όχι εξατομικευμένα και βλέπουμε αν όσοι ήρθαν με το ίδιο πλοίο είχαν την ίδια επαφή στη χώρα προέλευσης τους. Για πρώτη φορά κάνουμε τέτοιου είδους ανάλυση. μιλήσατε για προϋπολογισμό και πόρους, ας μην επαναλάβω αυτά που είπα στην αρχή, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Οι προσδοκίες είναι πολύ ψηλές και οι πόροι χαμηλοί σχετικά. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Σας ευχαριστώ και με συγχωρείτε αν τυχόν δεν απάντησα όλα τα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ πολύ Ρόμπερτ και αν δεν απάντησες κάποιο ερώτημα είναι μάλλον γιατί ε, εγώ σε πίεσα γιατί βλέπω ότι αναφέρθηκε σε έναν προς έναν σε όλους όσους έθεσαν κάποια ερώτηση. Έχουμε καθυστερήσει όμως πάρα πολύ και προσπάθησε να απαντήσει σε όλους. Ε, βλέπω και τις προτεραιότητές σας για το 2015 και θα ήθελα και πάλι να πω στα μέλη ότι η ουσία εδώ είναι ότι υπάρχει ε, ένα επιχειρησιακό πλαίσιο αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ε, προσδοκίες ε, για την ΕΑΣΟ, διότι πρέπει να προωθεί καλό άσυλο, διαδικασία λήψης αποφάσεων ε, και υπάρχουν μια σειρά από προσδοκίες, τις οποίες πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο να επιτύχουμε με βάση αυτούς τους πόρους που έχουμε. Ε, και τελικώς ε, η ΕΑΣΟ ε, προσφέρει αποτελέσματα. Και αυτό το οποίο λέμε σήμερα είναι ότι εμείς σε σχέση και με τη συζήτηση για την ετήσια έκθεση θα κάνουμε κάποιες προτάσεις με τους συντονιστές για να προχωρήσουν τα θέματα αυτά όχι μόνο για το κάθε θέμα μεμονωμένα το οποίο θα προκύψει το 2015 αλλά να έχουμε και κάποια απτά στοιχεία τα οποία έθιξαν οι συνάδελφοι. Θα τα αναφέρουμε αναλυτικά και θα προχωρήσουμε τις προτάσεις αναλόγως. Δεν θα πάει τίποτα χαμένο και βεβαίως θα επανέλθετε και για το, τις προτεραιότητες του 2015 και θα ακούσουμε ε, τι έχετε να μας πείτε. Διότι όπως βλέπετε υπάρχει σαφές ενδιαφέρον για το θέμα αυτό και σίγουρα πρέπει να υπάρχει και σχέση μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας εδώ σήμερα και για το γεγονός ότι δώσατε τόσο αναλυτικές απαντήσεις σε όλες μας τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Okay, colleagues, um, thank you. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Παρουσίαση από τον Πιέτρο Ρούσο, από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, ε, μια ειδική έκθεση, διότι τον Ιούνιο του 2010 ζητήθηκε μια έκθεση για τα διδάγματα που αντλήθηκαν για το σύστημα Σέγγεν ε, δεύτερη γενιά, το ΣΥΣ2. Ε, πρόσφατα η έκθεση του, δικαστηρίου, του ελεκτικού συνεδρίου, σας έχει διανεμηθεί. Έγινε μια συζήτηση ε, για το θέμα αυτό και η Μόνικα Χολμάγερ ε, ετοιμάζει μια έκθεση για τα όσα συζητήθηκαν στην Αρμόδια Επιτροπή και τώρα θα ήθελα να ε, ζητήσω από τον κύριο Ρούσο που είναι αποτελεκτικό Συνήδριο να μας παρουσιάσει την έκθεση και από εκεί και πέρα η κυρία Χολμάγερ θα πάρει το λόγο και θα μας πει κάποια πράγματα. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο και στον κύριο Κοέγιο ο οποίος είναι ο πρώην εισηγητής ε, για το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Πρώτα όμως να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ρούσο για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του. Κύριε Ρούσο. Μπορείτε να κάνετε την παρουσίασή σας και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων, κυρίες και κύριοι. La Cour des comptes européenne a publié Το ελεγκτικό συνέδριο στις 19 Μαΐου του 2014 δημοσίευσε μια ειδική έκθεση για τα διδάγματα που ατλήθηκαν από την ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν δεύτερης γενιάς, ε, το λεγόμενο SIS-2. Το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν, το SIS-2, χρησιμοποιείται από το 1995 από τους συνοριοφύλακες, τις αστυνομικές αρχές, ε, τις τελωνιακές αρχές και όσους είναι υπεύθυνου για τις θεωρήσεις διαβατηρίου στο χώρο Σέγγεν. Περιλαμβάνει πληροφορίες οι οποίες ονομάζονται σήματα ε, για άτομα τα οποία πιθανόν να εμπλέκονται σε σοβαρά εγκλήματα και υπάρχουν υποψίες ότι δεν έχουν την ε, δυνατότητα να ε, εισέλθουν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης περιλαμβάνει και λεγόμενα σήματα για εξαφανιστέντες και για ε, κλαπέντα ή απολεσθέντα αντικείμενα. Το 2001 το Συμβούλιο αποφάσισε να αντικαταστήσει το σύστημα αυτό από ένα σύστημα δεύτερης γενεάς, το SIS-2, το οποίο ε, ανέλαβε να αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο βασικός λόγος για την ανάπτυξη του ΣΥΣ2 ήταν για να επιτρέψει στα νέα κράτη-μέλη να διασυνδεθούν στο σύστημα. Επίσης ε, προβλέπεται το ΣΥΣ2 να περιλαμβάνει και τις ε, πιο προηγμένες τεχνολογίες και κάποιες επιπλέον λειτουργίες το ε, ελεγκτικό συνέδριο εξέτασε γιατί δεν δόθηκε το ΣΥΣ2 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια των αρχικών προθεσμιών. Και επίσης το ελεγκτικό συνέδριο εξέτασε κατά πόσον αντλήθηκαν κάποια διδάγματα από την διαχείριση του συστήματος και αν είχαν εφαρμοστεί και θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν έκανε έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων ε, για να αξιολογήσει κατά πόσο είναι ποιοτικά αυτά τα συστήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έδωσε το αρχικό σύστημα με πάνω από 6 χρόνια καθυστέρηση και με πολύ ε, μεγαλύτερο κόστο από, από αυτό το οποίο είχε εκτιμηθεί αρχικώς. Επίσης αξιολογήθηκε το πλαίσιο της διακυβέρνησης, ε, το οποίο δεν επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διορθώσει τα επιχειρησιακά συστήματα, καθώς επίσης και κάποιες αδυναμίες οι οποίες ήταν εις βάρος της διαχείρισης του προγράμματος ε, και κυρίως ε, κατά το πρώτο τμήμα της εφαρμογής μέχρι το 2009. Πιο συγκεκριμένα, οι αρχικέ προθεσμίε που είχαν καθοριστεί για το πρόγραμμα δεν ήταν καθόλου ρεαλιστικέ και η ανάπτυξη του προγραμματο συς ΣΥΣ2 ε, είχε προβλήματα αρχικής τελοποίησης ε, και ε, αντιμετωπίστηκαν προβλήματα εντό Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σύστημα εξελίχθηκε στη διάρκεια του προγράμματο ώστε να μπορεί να ανταποκραθεί στις ανάγκε των χρηστών και δεν ήταν επαρκώς σταθερό πριν από το 2010 το πέρασμα στο τελικό στάδιο έγινε τότε. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι το σύστημα το οποίο λειτουργεί σήμερα έχει πολύ καλύτερες δυνατότητες από αυτές που είχαν προβλεφθεί το 2001. Το ΣΥΣ2 διαθέτει ένα κεντρικό σύστημα το οποίο έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης και εθνικά συστήματα τα οποία έχουν αναπτύξει οι χώρες που συμμετέχουν στο χώρο Σέγγεν. Οι αρχικές εκτιμήσεις του κόστους του κεντρικού συστήματος ε, για τον ε, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ε, ήταν ε, πολύ κάτω των ε, ε, τελικών απαιτήσεων για επένδυση. Το συνολικό κόστος του ΣΥΣ2 έφτασε περίπου στις 500.000, 189.000 και πάνω από 330.000 ευρώ για τα εθνικά συστήματα. Και επιπλέον το βασικό, τα βασικά πλεονεκτήματα του ΣΥΣ2 έπαψαν να έχουν ενδιαφέρον που ήταν ουσιαστικά η εφαρμογή και η επέκταση του ΣΥΣΕΝΑ στις χώρες που εντάχθηκαν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το 2004 και το 2007. Επομένως, δεν έγινε εις βάθος ε, ανάλυση από πλευράς ελεγκτικού συνεδρίου της ε, ε, αποδοτικότητας του προγράμματος. Παρ' όλα αυτά αντλήθηκαν κάποια διδάγματα από την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος. Μπορέσαμε να αλλάξουμε προσέγγιση για το τελικό στάδιο το οποίο ξεκίνησε το 2010 και να εξοπλιστεί και να παρα, το συς με νέα στοιχεία και να, δοθεί το 2000, να παραδοθεί το 2013. Επίσης μπορούν να προχωρήσουν ε, και άλλα πολύ μεγάλα προγράμματα ε, πληροφορικής, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα των εφιών συνόρων. Το ελεγκτικό συνέδριο έδωσε αρκετέ συστάσει βάσει των παρατηρητερών σου για τη διαχείριση και ανάπτυξη του συστήματο πληροφορική ε, μεγάλη κλίμακα, τα οποία θα πρέπει να προσέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα και είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω στι ερωτήσει σα. Thank you very much. Um, Ευχαριστούμε πολύ. Η Μόνικα είναι εδώ. Τι κάνετε εκεί ψηλό κουβέντα έχετε πιάσει. Προσέχουμε στο μάθημα. Θέλετε να πείτε εν κάτι τώρα. Κάρλος. Εσύ πρώτος κύριος Κόλλιο ήταν ε, πρώην ε, εισηγητής, η ε, κυρία Χολμαϊρ εκεί πέρα που μιλούσε με το διπλανό της επίσης. Κύριε Κόλλιο, θέλω να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, πολύ καλή έκθεση και τονίζει τα προβλήματα που είχαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση με το σύστημα αυτό, με τις τεράστιες καθυστερήσεις και τα πολλά λεφτά που ψοδέψαμε. Τρία σχόλια θα ήθελα εγώ να κάνω. Τι πρέπει να κάνουμε, τι δεν πρέπει να κάνουμε και ε, τι έχουμε κερδίσει από αυτή τη διαδικασία. Πρώτον, τι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω πρέπει να αναγνωρίσουμε πως είχε δίκιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ασκούμε κριτική στην Κομισιόν για τη διαχείριση του συστήματος. Ζητάμε από το ελεγκτικό συνέδριο να κάνει τον έλεγχο και το συμπέρασμα απέδειξε πως είχαμε δίκιο. Δεύτερον, νομίζω πως πρέπει να διδαχτούμε από τα λάθη μας και να μην ε, κάνουμε τα ίδια λάθη και ε, ελπίζω να αντλήσαμε τα διδάγματα που έπρεπε. Και τέλος στο μέλλον πρέπει να ε, διαλέγουμε καλύτερα τις επιχειρήσεις με τις οποίες κάνουμε συμβόλαια. Δεν είχαμε νομίζω την σωστή ε, κρίση που θα έπρεπε και βεβαίως πρέπει να, εργαζόμαστε, να συνεργαζόμαστε με όλους. Δηλαδή, στην αρχή η Κομισιόν να συνεργαζόταν με τα κράτη-μέλη. Και συνειδητοποιούμε τώρα, μόνο αφού δημιουργήσαμε ένα διοικητικό συμβούλιο με τα κράτη-μέλη, πώς πραγματικά γίνεται η δουλειά και οριστικοποιείται το σύστημα. Δεύτερο σχόλιο. Τι δεν πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να συγχέουμε το SIS 2 και τη διαχείριση της Κομισιόν. Δηλαδή ήταν λανθασμένη η διαχείριση αλλά το SIS2 πρέπει να συνεχίσουμε να το στηρίζουμε, το χρειαζόμαστε για να έχουμε πιο ασφαλή σύνορα και οπωσδήποτε είναι ένα καλό έργο. Δεύτερον, όπως απέδειξε το ελεγκτικό συνέδριο, στο μέλλον δεν πρέπει να έχουμε προκήρυξη διαγωνισμού πριν να έχουμε αποφασίσει για τα πάντα. Το είπα αυτό χτες. Γιατί η πρώτη προκήρυξη έγινε πριν αποφασίσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Δεν έχει νόημα να αρχίσουμε να φτιάχνουμε ένα τεράστιο σύστημα χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι ε, νομικές απαιτήσεις. Δεν περίμεναν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να αποφασίσουν ε, τι θέλουν να κάνει το σύστημα. και πρέπει, όπως είπα, να αποφασίσουμε άρα εκ των προτέρων τι θέμε, τι χρειαζόμαστε. Και, όπως είπα, τι θέλουμε από αυτό το σύστημα. Ε, καμιά φορά δεν είναι εύκολο να επιβάλλουμε τέλη στους ε, αναδόχους γιατί οι ανάδοχοι θα μας πούνε μα, μα ζητάτε καινούργια πράγματα και μας ζητάτε καινούργια πράγματα κάθε μήνα ή κάθε τρεις μήνες. Τέλος. Πού καταλήξαμε. Ξέρουμε τι δεν πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Εν πάση περιπτώσει, το SIS2 είναι ένα καλό εργαλείο, όπως αναγνωρίζουν όλοι. Αστυνομία, δικαστική συνεργασία κτλ έχουμε ευρωπαϊκό SIS και παλέψαμε γι' αυτό και άρα όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να αξιολογούν την διαχείριση τώρα θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγε να γίνει έλεγχος προσωπικών δεδομένων στο SIS. δεν μπορούσε η υπηρεσία να μπει στο κτίριο γιατί δεν ήταν ευρωπαϊκό, ήταν υπό την επίβλεψη των γαλλικών αρχών. Και ε, δεν επετράπησε στι ευρωπαϊκές αρχές να μπουν στο κτίριο. Τώρα μιλάμε για ευρωπαϊκό όργανο. Έχουμε την νέα Λίζα τώρα, δηλαδή Έχουμε δηλαδή τεχνική εμπειρογνωμοσύνη, έλεγχο επιτόπου, έχουμε δηλαδή ε, κάποια επιτυχία, ακόμα και με τεράστια καθυστέρηση. Αυτά και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κάρλος, αναλυτικότατος ο συνήθως. Κυρία Χολμάιρ έχει προετοιμάσει το έγγραφο εργασία από την Επιτροπή Οικονομικών. Οπότε, ε, την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, με συγχωρείτε. Θέλετε να πείτε κάποια πράγματα. Ναι. Ευχαρίστω. Εκτό αν θέλει να μιλήσει συνάδελφο. Όχι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Όταν μου επεσήμανε ο Κάρλος Κοέλιο πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα, αρχίσαμε να τα αναλύουμε και είδαμε πάρα πολλά προβληματικά σημεία και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεκτικό συνέδριο, τον κύριο Ρούσο και όλους τους άλλους ελεκτές για την εξαιρετική δουλειά τους. Μας δίνει μια καλή αφετηρία για το τι δεν επιτρέπεται να ξανασυμβεί στο μέλλον. Τα λάθη τα οποία έγιναν Ναι, μας λέτε πως ε, δεν είχαμε αρκετούς ειδικού. Ε, ο προγραμματισμός ενός τέτοιου μέσου το οποίο θα πρέπει να δικτυώνεται διεθνώς, ε, να έχουν διάφορη πρόσβαση ήταν κάτι το δύσκολο και υπήρχαν και υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας και ούτε η εταιρεία ούτε η Κομισιόν είχαν τις απαραίτητες δυνατότητες. Αυτό για το μέλλον σημαίνει πως ε, όταν μιλάμε παραδείγματο χάρη για τα έξυπνα σύνορα ή για άλλο έργο πληροφορικής να υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό εμπειρία να δούμε τα οικονομικά με τρόπο λογικό και να δούμε το τι θέλουν τα κράτη-μέλη όταν αποφασίζουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Δηλαδή αυτό σημαίνει πως ε, θα ξέρουμε από εδώ και μπρος τι να κάνουμε και κάτι άλλο. Όταν δεσμεύεται κάποιος σε πληροφοριακά συστήματα ε, προσπαθούμε να μην έχουμε μονοπωλιακές δομές. Και πρέπει να προσέχουμε στους διαγωνισμούς μας ε, να μην ε, είναι εραστεχνική προκήρυξη. Γιατί πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι συμβατό και διαφανές και να μην δεθούμε με έναν ανάδοχο στην αιωνιότητα. Γιατί τι εννοώ δηλαδή αν ε, συμβαστούμε πάρα πολύ με έναν ε, μετά δεν μπορούμε να βάλουμε άλλον γιατί πρέπει να ξανακάνει όλη τη δουλειά από την αρχή κτλ. Αυτό πρέπει να γίνει πιο σαφές από ότι ε, με το SIS 2. Γιατί, γιατί με κάθε λάθος μας έβγαζε περισσότερα η εταιρεία. Και ε, ε, Βεβαίω, εντάξει, τώρα μειώθηκαν αυτές οι, οι αλλά το SIS 2 είναι ένα σημαντικό, αναγκαίο πρόγραμμα και καλό είναι ε, το ότι γίνεται στην Ευρώπη. Αλλά σε τέτοια προγράμματα πραγματικά πρέπει να έχουμε καλό προγραμματισμό από την αρχή και αυτοί οι οποίοι το κάνουν μετά να γνωρίζουν από την αρχή τι κάνουν και γιατί το κάνουν. Αλλιώς χάνουμε χρόνο και χρήμα και ασφάλεια. Σας ευχαριστώ. Δύο βουλευτές θα ακούσουμε και μετά θα τελειώσει ο κατάλογος. Κουτσίνη και Εμιλία. Η κυρία Κουτσίνη πρώτα. Κελίτσι, sorry. Βλέπω το όνομά σα σωστά συνέχεια. Ζητώ συγγνώμη, όμω δεν καταφέρνω να το προφέρω σωστά. Ξέρω, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι λίγο δύσκολο το επιθετό μου, δεν πειράζει. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν πρέπει να ε, το κάνουμε αυτό. Πρέπει όλοι να προφέρουμε τα ονόματα σωστά και το δικό μου προφέρεται ζήτερα και εγώ ζητώ συγγνώμη. Όχι, όχι, μην ανησυχείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Ρούσο, ο οποίος ε, μας παρουσίασε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για την ε, ε, περαιτέρω εξέταση που ζητήθηκε για το πρόγραμμα ΣΥΣ2. Ε, Δικαίω είναι επικριτική έκθεση, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι ταυτόχρονα είναι και ρισορροπημένη, διότι μας δίνει αντικειμενικά στοιχεία και μας ε, δείχνει σαφέστατα ε, όλους τους λόγους που οδήγησαν σε καθυστερήσεις και το λόγο για τον οποίο αυξήθηκε πραγματικά θεαματικά το κόστος και ήταν πολύ περισσότερο από αυτό το οποίο είχε προβλεφθεί αρχικά. Θα πρέπει επίσης να ευχαριστήσω και τους δύο συναδέλφους που μίλησαν πριν από μένα, κυρίως την εισηγήτρια στην Επιτροπή Ελέγχου του του που έκανε εξαιρετική δουλειά και κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα τα οποία πραγματικά θεωρώ ότι είναι ε, πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα. Η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου εξέτασε την ε, κατάλληλη χρήση και λειτουργία του συστήματος SIS-2 ε, και μας παρουσίασε μία σειρά από αίτια τα οποία οδήγησαν στην πολύ μεγάλη καθυστέρηση και στην πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των δαπανών. Ξεκινώντας από το αρχικό σφάλμα στην ανάθεση του έργου, διότι εκεί διαπιστώθηκε ότι θα ήταν λιγότερο δαπανηρή η επιλογή ε, η οποία κέρδισε το μειοδοτικό διαγωνισμό, που τελικώς αποδείχθηκε ότι κάθε άλλο ε, παρά τέτοια ήταν, όπως μας απέδειξε το ελεγκτικό συνέδριο, και επίσης υπήρχαν και μια σειρά από και δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίστηκαν κατά την εφαρμογή του συστήματος. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι οι επικρίσεις ε, ναι μεν ε, δεν μπορούν να αμφισβητήσουν την ανάγκη να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα ε, πληροφορική, το οποίο θα είναι πολύ προηγμένο και θα είναι στη θέση, η διάθεση τη αστυνομία των συνοριοφυλάκων, των τελωνιακών αρχών, ε, ε, για να μπορέσουν να γίνουν κατάλληλο έλεγχο των συνόρων. Και χαιρόμαστε που εφαρμόστηκε πλήρω το σύστημα στι 2 τον Απρίλιο του 2003 και που αντλήθηκαν διδάγματα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την εμπειρία αυτή με ένα κατάλληλο πλαίσιο διαχείρισης και διακυβέρνησης των ε, μεγάλων έργων πληροφορικής. Θα πρέπει βέβαια να επισημάνουμε ότι οι απαιτήσει των συστημάτων που θα πρέπει να αναπτύσσονται θα πρέπει να καθορίζονται εκ των προτέρων πριν ξεκινήσει το πληροφοριακό σύστημα. Και κάτι ακόμα πιο γενικό, αν μου επιτρέπετε, το γεγονός ότι Ζητήθηκε να εξεταστεί περαιτέρω ε, το θέμα αυτό και το γεγονός ότι έκανε τόσο καλή δουλειά το ελεγκτικό συνέδριο ε, έχει για μένα και μία πιο γενικού χαρακτήρα ε, καλή διάσταση διότι ζητάμε από όλα τα θεσμικά όργανα να διασφαλίσουν ότι θα γίνεται σωστή και καλή χρήση των δημοσίων πόρων. Ευχαριστώ πολύ. Η Κορνίλια. Κοιτάξτε, ειλικρινά, ένα τέτοιο έργο σε μια πόλη όπως η Δρέσδη είχαμε και εμείς κάτι ανάλογο. Δηλαδή η εκτίμηση του κόστου στην αρχή ήταν τελείως λανθασμένη και το αποτέλεσμα ήταν πως το τελικό κόστος ήταν εξαπλάσιο και Ε, το αποτέλεσμα ήταν πως οι υπεύθυνοι του έργου απολύθηκαν. Έτσι είναι το σωστό. Έτσι. Και όταν υπάρχει τόσο ε, επικριτική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για την οποία σας ευχαριστώ και βλέπουμε αυτό τον ερασιτεχνισμό πραγματικά, ε, δεν είναι δυνατό να μην υπάρχουν συνέπειες Οπότε η εκτίμηση αυτή του κόστους έγινε έτσι, ότι τους κατέβηκε. Έτσι κάθισαν σε ένα τραπέζι και είπανε, ξέρω εγώ να, πούμε ένα νούμερο. δεν είναι πτέσμα λοιπόν αυτό το οποίο συνέβη εδώ πέρα. Μιλάμε για ένα μεγάλο έργο το οποίο κόστησε 8 φορές παραπάνω από το προϋπολογισμένο. Ε, είναι σκάνδαλο. Τα ερωτήματα που θα ήθελα να πω, να κάνω τα εξή. Κάνατε συστάσεις ε, Εάν είχατε λοιπόν ε, ένα πράγμα να μας πείτε, ποιο θα ήταν το σημαντικότερο, η σημαντικότερη σύσταση προς την Κομισιόν και προς τους υπόλοιπους. Πείτε μας, σας παρακαλώ κάτι. Και θεωρείτε πως με τα διδάγματα αυτά πράγματι έγινε κανείς σοφότερος ή από το ένα μπαίνουν και από το άλλο βγαίνουν. Το ένα Σας ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα την Κομισιόν και μετά θα τελειώσουμε εδώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν εξ ονόματος Κομισιόν θα ευχαριστήσω και όσο και το ελεκτικό συνέδριο για την εξαιρετική του έκθεση και την κυρία Χολμάγερ για το κείμενο έγγραφο εργασίας της. Από ό,τι κατάλαβα δεν θέλετε πολύ εκτενώς τη θέση της Κομισιόν αλλά ευτυχώς τα έχουμε υποβάλει όλα αυτά γραπτά τα σχόλια μας μαζί με τα δικά σας προς την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά θα ήθελα να τονίσω μερικά στο παρελθόν έγιναν λάθη και η Κομισιόν δέχεται όλες τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Ταυτόχρονα όμως αναφέραμε περιπτώσεις όπου πιστεύουμε ότι η ανάλυση του δεν είναι πλήρης ιδιαίτερα ως προς το ρόλο του Συμβουλίου συνθήκες υπό τις οποίες εγγράφηκε αυτή η έκθεση πρέπει να τονιστούν. Το Συμβούλιο αποφάσισε να εφαρμόσει το ISIS 2, το SIS 2, χωρίς πρόταση της Κομισιόν ούτε σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Και μερικά όσα ζητούσε η έκθεση στην αρχή δεν προβλεπόταν. Στην αρχή Θέλαμε απλώς να συνδεθεί το σύστημα με τη, τα συστήματα των χωρών που εφαρμόζουν το Σέγγεν. Με τον καιρό προσθέθηκαν και νέα αιτήματα, τεχνικά στοιχεία, προδιαγραφές χρειάστηκαν να αλλάξουν και προφανώς αυτό είχε επιπτώσεις και στο χρονοδιάγραμμά του και στην κοστολόγησή του. Είναι πολύ απλοϊκό να λέμε ότι το ΣΥΣ κόστισε 8 φορές παραπάνω από ό,τι προβλεπόταν και ότι αυτό είναι σκανδαλώδες. Εντάξει, ήταν η διαδικασία λίγο περίεργη, αλλά δεν ευθύνεται η Κομισιόν γι' αυτό. Αν θέλουμε να πάρουμε μαθήματα, αν θέλετε να πάρετε μαθήματα, πρέπει τότε να δείτε και το πώς δημιουργήθηκε, πώς γεννήθηκε αυτό το σχέδιο. Ακούστηκαν δηλώσεις για έλλειψη διαφάνειας της Κομισιόν Πάλι δεν έχω το χρόνο να σας τα πω λεπτομερώς, αλλά στα γραπτά μου σχόλια βλέπετε ότι πρόκειται για παρεξήγηση για να το πω έτσι. Η Κομισιόν πάντοτε ήταν διαφανέστατη για τις, τους διαγωνισμούς. Δεν μπορούμε να τα δεχτούμε αυτά τα λόγια. Ήμασταν πάντοτε επαγγελματικότατοι στην εφαρμογή των κανόνων στην εφαρμογή των δημοσιονομικών κανονισμών και στην υποβολή των προγραμμάτων μας στον έλεγχο των δημοσιονομικών αρχών. Δεν έχουμε κανένα λόγο να, κάνουμε, να ακούμε τέτοιες κατηγορίες. Τέλος κύριε Πρόεδρε, για το μέλλον, σήμερα έχουμε το ΣΥΣ2 που είναι πολύ αποτελεσματικό και από τότε που τέθηκε σε ισχύ πριν από 9 μήνες 1,3 δισεκατομμύρια όχι λιγότερα προσβάσεις έγιναν στο σύστημα από αρχές των χωρών μελών 86.000 προσβάσεις για έρευνα και προειδοποίηση και το ΣΥΣ2 γενικά είναι πολύ βοηθητικό. Βοηθάει τις κυβερνήσεις πολύ αποτελεσματικά. Και ελπίζουμε να συνεχίσει και στο μέλλον. Άλλο για το μέλλον, τα μαθήματα που πήραμε για άλλα ηλεκτρονικά προγράμματα όπως τα έξυπνα σύνορα. Εδώ μπορώ να σας, να σας βεβαιώσω ότι δεν άρχισαν διαγωνισμοί χωρίς να έχει προηγουμένως πλήρως ολοκληρωθεί η νομοθεσία. Αυτό ήταν ένα από τα μαθήματα που πήραμε. Η προετοιμασία των εξύπνων συνόρων θα συμπεριλαμβάνει την Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ισότιμα. Πήραμε μαθήματα λοιπόν από το παρελθόν και θεωρούμε ότι γι' αυτόν τον λόγο η έκθεση αυτή θα μας βοηθήσει για καλύτερη διευθέτηση στην Ένωση και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταία συντομότατα συμπεράσματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ, πολύ σύντομα. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω, διότι αυτά τα οποία ακούστηκαν γενικά και είμαι πολύ ικανοποιημένο διότι όλα τα μέλη αναγνώρισαν ε, το διεξοδικό έργο του ελεγκτικού συνεδρίου, την ισορροπία του και την ευστοχία των όσων ε, πρότεινε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ελεκτές μας. Ε, αν με επιτρέπει ο κύριος Πρόεδρος, πολύ σύντομα θα ήθελα να παρέμβω μόνο για το ερώτημα της κυρίας, ε, της οποίας ε, δυστυχώς δεν θυμάμαι πολύ καλά το όνομα ε, και ζητώ συγγνώμη, που ρώτησε ποιες ήταν οι συγκεκριμένες συστάσεις του Συμβουλίου και πώς λειτουργεί το θέμα αυτό. Η η σύσταση νομίζω είναι η δεύτερη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα πληροφοριακά ε, προγράμματα μεγάλης κλίμακας ε, στην κατάλληλη προετοιμασία. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική σύσταση, ε, διότι είναι πάρα πολλά τα λάθη σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση και η σύσταση φαίνεται ότι είναι αυτονόητη, αλλά είναι πολύ σημαντικό να την αναφέρουμε. Κατά τα λοιπά, εμείς ε, για την παρακολούθηση της έκθεσης αυτής ε, θα συνεχίσουμε. Προς το παρόν το ελεγκτορικό συνέδριο ε, σταματάει στον έλεγχο που έκανε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δέχεται τις συστάσεις και θα κάνει και ανακοινώσεις από αυτού. Ευπρόσδεκτα αυτά και να σας πω ότι αν γίνει παρακολούθηση στη συνέχεια, κατόπιν ετήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της έκθεσης αυτής, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ κύριε Ρούσο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και συγγνώμη που σας πίεσα να βιαστείτε εδώ στο τέλος. Σας είμαστε ευγνώμονες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, um, Αγαπητοί συνάδελφοι, καθυστερήσαμε λίγο. Να προχωρήσουμε λοιπόν πολύ γρήγορα στο επόμενο σημείο. Σημείο 6. Παρουσίαση της νομικής υπηρεσίας για την προδικαστική απόφαση του Irish High Court ε, ε, γνωρίζουν οι συνάδελφοι περί τίνος πρότυχητε, επομένως θα περάσω στην ουσία. Πρόκειται για μια απόφαση του ε, High Court of Ireland, αλλά μας ενδιαφέρει αυτό διότι έχουμε και την απόφαση για τον ασφαλή λιμένα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και κατά πόσον είναι απόλυτα δεσμευτικό το γεγονός ότι μια προστασία, ε, ε, υπηρεσία προστασίας δεδομένων μπορεί να ξεκινήσει ε, διαδικασία προστασίας βάσει του ασφαλούς λιμένα. Είναι πάρα πολύ σημαντική η απόφαση. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι η αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή και είναι η αρμόδια για τις ε, ε, υποθέσεις οι οποίες συζητούνται στο δικαστήριο, θα συζητήσει για το θέμα αυτό αύριο. Θα γίνει και κλεισμένον των θυρών και θα σας πω δύο λόγα γι' αυτό. Θα πω γι' αυτό σε μισό λεπτό η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και εδώ αναφέρομαι και στα νέα μέλη, τα οποία δεν είναι και τόσο εξοικειωμένα με την ε, νομοθεσία για τον ασφαλή λιμένα. Είναι πολύ σημαντικό όμως και ότι η Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών, αφού ακούσουμε και την νομική υπηρεσία γενικά για τον ασφαλή λιμένα, να συζητήσει το θέμα αυτό και κλεισμένο των θυρών, ε, γιατί έχουμε και τους ε, αρμόδιους υπουργούς που θα έρθουν εδώ. Ε, θα ήθελα λοιπόν να μην γίνει πλήρη συζήτηση μετά από την παρουσίαση της νομικής υπηρεσίας σήμερα, πριν συζητήσει το θέμα αυτό η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Υπάρχει το εξής βέβαια, η συζήτηση αυτή θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, ε, επειδή υπάρχουν και δικαστικές διαδικασίες και σχετίζονται αυτά και με τα έγγραφα τα οποία διανέμονται στα μέλη, τα οποία θα πρέπει να επιστραφούν στη γραμματεία, επομένως η συγκεκριμένη συνεδρίαση θα πρέπει να γίνει και κλεισμένο των θυρών. Θα ήθελα λοιπόν να γίνει συνεδρία συγκεκριμένα των θυρών, θα ε, δοθούν τα έγγραφα στα μέλη. Υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει κάτι διαδικαστικό, Σόφι, έχει κάτι διαδικαστικό να πεις. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, νομίζω ότι είναι κρίμα που ξεκινούμε τόσο καθυστερημένα. Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα, αλλά θα πρέπει να φύγω γιατί πρέπει να προεδρεύσω και εγώ σε κάποια συνεδρία σε ένα τέταρτο. Όσον αφορά το τμήμα του ε, γεγονότος ότι συνεδριάζουμε και κλεισμένο των θυρών, οι συνεδριάσεις κλειμένων των θυρών, από ό,τι έμαθα, δεν ηχογραφούνται. Επομένω δεν μπορούμε μετά να δούμε κατά πόσον είναι αιτιολογημένο να γίνει συνεδρίαση και κλεισμένο των θυρών. Εάν να δοθεί η δυνατότητα λοιπόν για συνεδρίαση και κλεισμένο των θυρών θα πρέπει να ηχογραφούνται, οπότε σε περίπτωση που αμφισβητεί κάποιο την απόφαση να μπορούμε να επαληθεύσουμε αν ήταν αιτιολογημένη ή όχι. Σόφι, πριν ε, απαντήσω υπάρχει κάτι ακόμα, αυτό. Συνάδελφοι, υπάρχουν κάποια άλλα ερωτήματα για το κατά πόσον θα πρέπει να γίνει και κλεισμένο των θυρών η συνεδρίαση και το ερώτημα της Σόφη. Κορνίλια, θέλεις και εσύ να το πεις τώρα για να απαντήσω και στα δύο. Ναι, ε, ως συνήθως είμαι κατά. Δεν είναι δυνατό να το συζητήσουμε και δεν είναι και ικανοποιητική η διαδικασία αυτή. Πρέπει τουλάχιστον εκ των προτέρων να υπάρχει μια αιτιολόγηση για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Μάλιστα, ευχαριστούμε Κορνιλία. Να τα απαντήσω και τα δύο. Πρώτα απ' όλα, εγώ το παίρνω πάρα πολύ σοβαρά αυτό το ζήτημα.